Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ και αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας με τις συνήθεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζω όλους και σας υπενθυμίζω ότι αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση αυτή και όσον αφορά την προτεραιότητα της διερμηνίας, αυτή δίνεται στις γλώσσες των τακτικών μελών της ε, ΣΕΝΤΕ της Υποπιτροπής μας. Η μερίσια διάταξη τώρα εγκρίνεται. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρείται εγκεκριμένη. Έχουμε τίποτα για πρακτικά. Όχι. Δεν έχουμε πρακτικά. Όσον αφορά ανακοινώσει τη Πρόεδρου τώρα, μία παρατήρηση έχω να κάνω, ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούμε με την ε, Γερμενίδα Ομοσπονδιακή Υπουργό Άμυνα, την κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λέιεν, η οποία θα έρθει στο Στρασβούργο την Τρίτη κατά πάσα πιθανότητα δύο με τρεις το μεσημέρι περίπου. Και θα συναντηθούμε μαζί της από κοινού με την Επιτροπή ΑΦΕΤ εξωτερικών υποθέσεων. Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στα ουσιώδη θέματα της ημερήσιας διάταξης και έχουμε Πρώτα απ' όλα το σχέδιο έκθεσης για τις εξαγωγές όπλων, εφαρμογή της κοινή θέσης 2008 κάθετος 944. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μποντήλ Βαλέρο. Συνεπώς, παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά, οπότε παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Εντάξει, είμαστε όλοι έτοιμοι. Ωραία. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που με εμπιστευτήκατε. Γιατί έτσι μπόρεσα να ασχοληθώ και πάλι με την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου. Και ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, ε, εξαγωγικών ε, συμβατικών όπλων, γιατί με βοήθησαν να συντάξω την έκθεση αυτή. Άκουσα δηλαδή την άποψη των εκπροσώπων των χωρών μελών και θα συναντηθώ μαζί τους, μαζί με τα μέλη της ΚΟΑΡ, με της ομάδας αυτής ε, για τις εξαγωγές συμβατικών όπλων, ξανά σύντομα. Συνεργάζομαι και με διάφορες ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Συναντήθηκα με εκπροσώπους της βιομηχανίας, της αμυντικής βιομηχανίας και έτσι μπόρεσα να ετοιμάσω και το σχέδιο εκθεσής μου. Μετά από την τελευταία έκθεση δεν έγιναν και πολλά. Ο πόλεμος στο Ιράκ και στη Συρία συνεχίζεται, δεν έχει τηθεί ακόμα το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, οι τρομοκράτες στην Ευρώπη μάλλον αυξάνονται αντί και υπάρχει μεγάλη πίεση γενικώ. Οι δημοσιογράφοι όλο και περισσότερο μα μιλούν για πωλήσει που γίνονται από χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Ενωμένο Βασίλειο, που δίνουν περισσότερες άδειε στη Σαουδική Αραβία, για εξαγωγέ στη Σαουδική Αραβία, μετά τον πόλεμο μάλιστα στην Ιεμένη. Και επίση υπάρχει και εξοπλισμός, αμυντικό όπλα ε, προ χώρε ε, οι οποίε κανονικά καλύπτονται με μπάρκο. Οπότε δεν τηρούνται πάντα τα κριτήρια όπως θα έπρεπε τα κριτήρια της κοινή θέση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυστηρά να τηρούνται τα κριτήρια αυτά. Είναι ζωτική σημασία αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την προστασία των ανθρώπων τόσο σε τρίτες χώρε όσο και στην Ευρώπη. Δεν έχουμε εγγύηση ότι τα όπλα τα οποία εξάγουμε δεν θα στραφούν εναντίον μας κάποια στιγμή. Εδώ, στη δικιά μας επικράτεια ή αλλού. Τα όπλα πολλούνται σήμερα παράνομα ενώ στην αρχή ήταν νόμιμα. Αυτή είναι μια απειλή σε βάρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο μακροπρόθεσμα και να έχουμε και μια αρχή πρόληψη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το δημοκρατικό έλεγχο επίσης, στην ε, σταθερότητα, την περιφερειακή, τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε φορά που αποφασίζουμε να πουλήσουμε όπλα σε μια χώρα. Επίσης, ο έλεγχος στις χώρες προορισμού πρέπει να βελτιωθεί. Χρειάζονται καλύτερες εκθέσεις, περισσότερη διαφάνεια και πρέπει να έχουμε πιο εύκολα πρόσβαση στις εκθέσεις κριτηρίων, πώς εφαρμόζονται δηλαδή τα κριτήρια αυτά. Οπότε σήμερα είμαι έτοιμη να συζητήσω μαζί σας για αυτό το θέμα. Ε, προσβλέπω και σε τροπολογίες, έτσι, από τους γεώδεις συζητητές και τους συναδέρφους γενικότερα. Θα δουλέψω πάνω σε αυτές τις τροπολογίες μαζί σας, προκειμένου να πετύχουμε όσο γίνεται ευρύτερη συνεργασία και να μπορέσουμε έτσι να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική λύση. Και εγώ θα υποβάλω τροπολογίες, ακριβώς επειδή χρειάστηκε να δουλέψω με μια συγκεκριμένη μορφή. Ε, το πρώτο μου σχέδιο είναι σύντομο, πιο σύντομο από ό,τι περίμενα. Θα υπάρξουν τεχνικές τροποποίησεις, δίχως άλλο στο κείμενο, προκειμένου αυτό να είναι πιο σαφές και ξεκάθαρο. Περιμένω τα σχόλιά σας τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος, για την παρουσίαση αυτή. Θέλω να επιθυμίσω στους συναδέρφους ότι είχαμε οργανώσει, η υποπιτροπή μας δηλαδή, και ένα εργαστήριο με εξαίρετους συμμετέχοντες. Ποιον έχουμε εδώ σκιώδη ηγητή. Αλλά προηγουμένως κάτι θέλει να προσθέσει η κυρία Βαλέρο. Να θέλω να κάνω μια παρατήρηση γιατί νομίζω ότι εγώ μίλησα για τη Συρία και από κάπου στη μετάφραση ακούστηκε κάτι για τη Βόρεια Κορία. Εγώ για Συρία μίλησα, λέει η κυρία Βαλέρο. Καλώς. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος ε, Τουνέλκεν Κέλλαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την συνάδελφο Μποντιλ Βαλέρο για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας, για την διαφάνεια, για το ανοιχτό της πνεύμα. Και για το γεγονός ότι ήταν ε, έτοιμη να βοηθήσει ώστε να λυθούν οι διαφορές μας. Συμφωνούμε λοιπόν ότι όντως υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό του ελέγχου εξαγωγών όπλων και οπλισμού. Και αυτό να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πιο αποτελεσματικό, γιατί τα βλέπουμε στη γειτονιά μας, πολύ κοντά μας, ε, σειράξεις, ένοπλες σειράξεις που οφείλονται στον ε, τεράστιο αριθμό εξαγωγών όπλων. Το να μιλάμε για κούρσα, για αγώνα εξαγωγών δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Πάντως, αυτό με το οποίο συμφωνώ είναι ότι χρειάζεται μια πιο ομοιόμορφη ερμηνεία των κριτηρίων, αξιολόγηση κινδύνου και βεβαίως διαφάνεια. Συνεπώς, με αυτά συμφωνούμε. Τώρα, ποια είναι η θέση του ΕΛΚ. Θέλουμε να ενισχυθεί το θέμα της αυτοάμυνας των χωρών μελών και τη σημασία που έχει η αμυντική μας βιομηχανία. Θα προτείνουμε διάφορες τροπολογίες από αυτού. Και θέλουμε και να υπογραμμίσουμε και την ε, τεχνολογία ως βιομηχανική βάση της ε, αμυντικής μας βιομηχανίας στα πλαίσια πάντα της ΚΕΠΑ. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι εμείς είμαστε περισσότερο υπέρ του να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων και όχι να τα επεκτείνουμε ή να επεκτείνουμε το εύρος εφαρμογής τους. Πιστεύω πάντως ότι μπορούμε από κοινού να προχωρήσουμε και να λάβουμε υπόψη μας διαφορετικές απόψεις οι οποίες τελικά στο κάτω-κάτω δεν είναι και τόσο διαφορετικές μεταξύ τους. Γιατί στο κάτω-κάτω όλους μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό της εξαγωγής όπλων που μερικές φορές καταλήγουν σε λάθος χέρια και μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την επέκταση των συγκρούσεων. Ευχαριστώ σε ευχαριστούμε. Η κυρία Γιάλα Σέντερ εκ μέρου των Σοσιαλιστών τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην κυρία Βαλέρο για το σχέδιο εκθεσή τη. Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε ε, διάφορα πράγματα, διάφορες ιδέες ε, δικές μας που διατυπώσαμε μέσα στο 2015 και εμείς με την προηγούμενη έκθεση όλο αυτό το θέμα με τον κατάλογο ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για παράνομες εξαγωγές ή έχουν συμμετάσχει σε παράνομες εξαγωγές εμπόριο όπλων και είναι καλό να την έχουμε, τον έχουμε υπόψη μας αυτό τον κατάλογο. Κατά τα άλλα και εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία ότι εκθετικά έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές όπλων και ακριβώς γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την εφαρμογή των κριτηριών. Μάλιστα εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να κοιτάμε μήπως μπορούμε να ενισχύσουμε ή να αυξήσουμε τα κριτήρια αυτά. Γιατί τώρα με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής, σε κάθε επίπεδο, ίντερνετ, black internet κτλ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν νέοι κίνδυνοι και άρα πρέπει να είμαστε σε θέση να βοηθούμε τις χώρες μέλη και τις κυβερνήσεις τους να έχουν αρκετούς πόρους για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο τουλάχιστον έχουν τις ίδιες δυνατότητες που έχουν και αυτοί που προβαίνουν στις παράνομες εξαγωγές να μπορούν και οι χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα με τα ίδια όπλα, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι επίσης πολύ σημαντικό, μια που φτάνουμε στον καθορισμό μιας ευρωπαϊκής επιτέλους πολιτικής άμυνας, Νομίζω ότι και στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να φροντίσουμε οι χώρες μέλη να συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους. Να βελτιωθεί επίσης η οικονομία κλίμακας. σε σχέση με τον αμυντικό ευρωπαϊκό εξοπλισμό, αλλά και όσον αφορά τις εξαγωγές, για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια δηλαδή, αυτό μας ενδιαφέρει και να μην υπάρχουν ε, τύχοι που να μην ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος ή άλλα να λέει άλλα να κάνει. Πρέπει λοιπόν να εμβαθύνουμε περισσότερο στις επιπτώσεις που θα έχει το Brexit σε, σε μια τέτοια ρύθμιση όπως είναι αυτός ο κανονισμός. Γι' αυτό και θα υποβάλουμε και τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μας, μας απασχολεί πολύ ήδη η συγγήτρια αναφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις εξαγωγές τους στη Σαουδική Αραβία. Χωρίς διαφάνεια για τις άδειες αυτές που έδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και στα πλαίσια του Brexit να έχουμε υπόψη μας αυτό το παράγοντα και να μην μειωθούν οι απαιτήσει που θα επιβάλλουμε σε σχέση με τόσες ισχύουν σήμερα απέναντι στον Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποιες τρίτες χώρες ακολουθούν τους ίδιους κανόνες της κοινής δεν θα έπρεπε να υπάρξει διαφοροποίηση, αντίθετα θα πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχο γιατί πολλά από αυτά που είπε η συγγήτρια είναι απολύτω σωστά και ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Χαβιέρ Νάρτ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το έργο της κυρίας Μποντήλ Βαλέρο είναι εξαίρετο και το λέω όχι για να την ευχαριστήσω, αλλά γιατί πραγματικά ισχύει. Εγώ δεν βλέπω να θέλω να τροποποιήσω κάτι σημαντικό. Όμως, πρώτα απ' όλα, πρέπει να έχουμε κυρώσεις αποτελεσματικές όταν παραβιάζονται τα οκτώ κριτήρια τα οποία έχουμε αποφασίσει στην κοινή θέση πρέπει ξεκάθαρα να λέμε ότι κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τηρούν τα κριτήρια αυτά. Άρα πρέπει να τονίσουμε την απέτησή μας να τηρούν τα κριτήρια αυτά, αλλιώς να υπάρχουν κυρώσεις. Φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να μηνθεί. Φυσικά και οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις ε, άμυνας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά να μέσα σε αυτό και την λαθροδιακίνηση όπλων, μέσω διόδων σκοτεινών ή μη παράνομων για να μπορεί κανείς τελικά να έχει κέρδος προσωπικό, όχι. Γι' αυτό λοιπόν να τηρούνται τα κριτήρια, αλλιώς να υπάρχουν αποτελεσματικές κυρώσεις. Μερικές φορές οι πληροφορίες είτε δεν έρχονται καθόλου από τις χώρες μέλη ή έρχονται πάρα πολύ αργά. Και αυτά πρέπει να τα λέμε με ειλικρίνεια. Δεύτερον, πρέπει να ζητήσουμε οι επιχειρήσεις ή οι ενδιάμεσοι εμποροί που παραβιάζουν τα 8 κριτήρια είτε να επιβάλλονται σε αυτούς τους κυρώσεις είτε ακόμα καλύτερα να λέμε ότι υπάρχει μια παράβαση και έτσι σταματάει η συνεργασία μαζί τους, τους βγάζουμε από τη μέση στο εμπόριο αυτό και να ξέρουν ότι δεν θα μπορούν πια να συμμετέχουν. Κάτι άλλο αποφασιστική σημασία είναι το εξή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε άδειε με τις οποίες κατασκευάζονται όπλα σε τρίτες χώρες με τεχνολογία της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Δεν ε, τα ξέρω βέβαια πολύ καλά, αλλά είναι γνωστό ότι μέσα από τρίτες επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται ευρωπαϊκή τεχνολογία και με αυτήν δημιουργούνται όπλα τα οποία στη συνέχεια όμως εξάγονται χωρίς περιορισμό. Δεν είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιούμε την κοινή λογική και να αφήνουμε τη δικιά μας τεχνολογία να βοηθάει να κατασκευάζονται όπλα αλλού, τα οποία τελικά καταλήγουν ούτε ξέρουμε πού. Συνεπώ, η τεχνολογία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιαδήποτε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγεται σε τρίτη χώρα, πρέπει να υποβάλλεται στου ίδιου περιορισμού όπως και όταν η παραγωγή γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς έχουμε μια μαύρη τρύπα εδώ, μέσα από την οποία αυτό το εμπόριο του θανάτου εξακολουθεί να λειτουργεί. Και τελειώνω με το εξή. Οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις ασφάλειας είναι αναπόφευτες. εξαιτίας μιας πολιτικής εξωτερήκευσης αυτού που δεν θα έπρεπε να εξωτερικεύεται, που είναι η ασφάλεια και η άμυνα. Για λόγους όμως προπολογισμού το κάνουμε ή και για λόγους αισθητικής θα έλεγα, γιατί θεωρούμε ότι είναι καλύτερα να γίνονται εκπτώσεις στις ιδιωτικές εξωτερικές υπηρεσίες ασφάλειας παρά ε, στη δικιά μας, δημόσια στο δικό μας στρατό ή τη δικιά μας αστυνομία για παράδειγμα. Όμως αν είναι κάποιος ο οποίος δουλεύει σε τέτοιες επιχειρήσεις, πρέπει να ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι καθαρές, ότι δεν γίνονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παράδειγμα. Και αν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε δεν πρέπει να παίρνουν όπλα επιχειρήσεις αυτές. Εγώ δεν είμαι υπέρ της υποκρισίας, είμαι υπέρ του ρεαλισμού. Και τις αρχές μας να τις στηρούμε πραγματικά. Η πρόεδρος, η κυρία Λούζινγκ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε η συνάδελφος. Είμαστε πάλι εδώ, τόσα χρόνια αργότερα, λέμε τα ίδια πράγματα και συμφωνούμε. Είναι πολύ ανησυχητική αυτή η κατάσταση. Νομίζω πως Βλέπουμε πως συμφωνούμε όλα αυτά τα χρόνια, επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, υπάρχουν εξαγωγές σε περιοχές επικίνδυνες και ας χρησιμοποιήσουμε τη σωστή έκφραση σε περιοχές ε, που υπάρχουν εμπόλεμες σειράξεις. Υπάρχει υπάρχουν πάλι τα ίδια, βλέπουμε πάλι να μιλάμε για ανάπτυξη, βλέπουμε πάλι πώς οδηγούμαστε στα ίδια συμπεράσματα, χρησιμοποιούμε αυτά τα 8 κριτήρια. Σημαντικό είναι ε, να γνωρίζουμε ότι αυτά τα 8 κριτήρια είναι κριτήρια που δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Η συγγήτρια μας ε, παρουσίασε μία έκθεση η οποία συμπεριλαμβάνει αρκετά από τα στοιχεία που ήθελε να συμπεριληφθούν η ομάδα μου. Και εμείς έχουμε παρόμοιες ε, απαιτήσει από την έκθεση αυτή. Και σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, να πω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα αυτό. Και να μην θεωρούμε ότι είναι το ίδιο τα παράνομα και τα, και τα απαγορευμένα είδη. Είναι, πιστεύω λοιπόν, σωστό να είναι πιο αυστηρέ οι κυρώσει και να είμαστε κι εμείς πολύ πιο αυστηροί με τη χορήγηση αδειών. Οι άδειε αυτέ θα πρέπει να χορηγούνται από ε, τα κράτη, αλλά κοιτάξτε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε μάλλον τόσε άδειε στη Σαουδική Αραβία που η κατάσταση ε, έχει ενταθεί πάρα πολύ. Σίγουρα οι λόγοι είναι οικονομικοί, έχουν σκοπό το κέρδος, εμπλέκονται πολύ κλάδοι της βιομηχανίας της εξαγωγής όπλων, αλλά πρέπει να δούμε τι είναι σημαντικό εδώ. Μετά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες ε, οι οποίες ε, έχουν άδειες, αλλά υπάρχουν γεωπολιτικές πολιτική και γεωστρατηγική ε, λόγοι. Γι' αυτό είναι, έχουν φιλικές σχέσεις με κάποια άλλα κράτη. Ε, η Γερμανία, για παράδειγμα, θεωρεί τη Σαουδική Αραβία πολύ σημαντικό στρατηγικό εταίρο. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει τι κάνουν αυτές οι χώρες με τα όπλα που τους ε, πουλούν σε άλλες χώρες στον κόσμο. Νομίζω πρέπει να αναφερθούμε λοιπόν σε αυτή τη γεωστρατηγική διάσταση. Μετά, Νομίζω πως υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις ε, σε ό,τι αφορά την πίεση που πρέπει να ασχηθεί σε ορισμενα και στις κυρώσεις. Και φυσικά ξέρουμε όλοι πως οι στόχοι είναι δεσμευτικοί. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ παράλογο ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε τις κυρώσεις και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Μετά, ε, υπάρχουν και πολλά σημεία στα οποία πιστεύω πως μπορεί να βελτιωθεί η έκθεση και γι' αυτά θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Αναγκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Μποντήλ Βαλέρο για την πολύ σημαντική η έκθεση, είναι περιεκτική, έχει συγκεκριμένες προτάσεις, κάνει μια λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης. Να αναφερθώ σε, στην εθελοντική, στον θελοντικό χαρακτήρα της τάσης που είχαμε μιλήσει όλα το 2008. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας το 2009 αυτή έγινε μια κοινή θέση για όλα τα κράτη-μέλη. Φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε και να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δέσμευση και επίπεδα εφαρμογή από κράτο μέλο σε κράτο μέλο και νομίζω πω υπάρχει μια γενικότερη επιδείνωση τη κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Αυτό τουλάχιστον ε, αναφέρει η έκθεση, η ετήσια έκθεση των τελευταίων δύο ετών. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αντί να επιληθούν έχουν επιδεινωθεί και αυτό διότι υπάρχουν σε διάφορα κράτη-μέλη διάφορες οντότητες οι οποίες ε, εκδίδουν άδειε για εξαγωγή όπλων και δεν δέχτηκαν όλες να δώσουν στοιχεία. Όταν προσπαθούσαμε να συντάξουμε την ετήσια έκθεση και αυτό το διαπίστωσα και η διεισόμαση. Κάποια στοιχεία περνούσαν πρώτα από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετά συμπεριλαμβάνονταν στην ετήσια έκθεση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ε, εταιριών οι οποίοι έκαναν εξαγωγές χώρες οι οποίες θα έπρεπε να είναι αποκλεισμένες από τις εξαγωγές σύμφωνα με την ε, κοινή θέση της Ένωσης. Μετά στην έκθεση αναφέρονται αρκετά σωστά θεωρώ σημεία και να πω πως είναι απαράδεκτο δεδομένων των απειλών που ακούγονται και κάποιες απειλέ δεν μένουν μόνο στα λόγια, είναι πραγματικές επιθέσεις οι οποίες γίνονται ει βάρο Ευρωπαίων πολιτών. Συμπεριλαμβάνω και τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες αυτές ε, επιθέσεις συνδέονται με την έλλειψη ελέγχου στις εξαγωγές όπλων. Όλοι γνωρίζουμε πλέον πώς έγιναν οι επιθέσεις στο Παρίσι και πόσο εύκολο ήταν να αγοράσουν όπλα από το Βέλγιο οι τρομοκράτες. Με λίγες χιλιάδες ευρώ που ένα αυτόματο. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο να μην τηρείται η κοινή θέση από όλα τα κράτη-μέλη. Και πρέπει να τονιστεί αυτό έντονα στην έκθεση και να παροτρύνουμε την Επιτροπή να δράσει. Διότι η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να δράσει, είναι μια δεσμευτική κοινή θέση για όλα τα κράτη-μέλη. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, γίνονται εξαγωγές όπλων στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα η οποία ξεκάθαρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Ε, μια χώρα η οποία δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ιεμένη, προκαλεί ένοπλες σειράξεις. Τις στηρίζει. Αυτός δεν είναι εταίρος μας στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και στην προσπάθεια για παγκόσμια ασφάλεια. Γι' αυτό συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες των συναδέλφων ε, για τις ε, τεχνολογίες, για παράδειγμα για τα οπλισμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη. Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί εντόνως τους ε, εμπειρογνώμονες και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης με ανησυχεί πάρα πολύ η έλλειψη ελέγχου σε άλλες εξαγωγές τεχνολογικών προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πόλεμο, στα είδη διπλής χρήσης που στόχο έχουν την καταστολή και την παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων σε πολλές χώρες. Θεωρώ λοιπόν πως είναι μια πολύ σημαντική έκθεση και το Κοινοβούλιο θα βοηθούσε πάρα πολύ την κατάσταση ασφαλείας εάν υιοθετούσε μια πολύ σκληρή, αυστηρή στάση και κατονομάσει τις χώρες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Δηλαδή τις τρεις χώρες που εξάγουν όπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο που δεν έχουν υποβάλει λεπτομερείς καταλόγους εξαγωγών, γιατί ακριβώς υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό. Ευχαριστώ. κύριος Γκάλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στις παραγράφου ε, παραγράφους 13 και 14. Εκεί να εστιάσω την προσοχή μου. Γιατί εκεί πρόκειται για την προαγωγή ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όσοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις στα διάφορα κράτη καλούνται να αποφασίσουν κατά πόσον θα εγκρίνουν ένα αίτημα για εξαγωγές ή όχι. Αυτοί λοιπόν γνωρίζουν πολύ καλύτερα περί τίνος πρόκειται ή θα είναι σε καλύτερη θέση να λάβουν τη σωστή απόφαση αν έχουν ε, όχι μόνο τις εθνικές ε, πληροφορίες αλλά πληροφορίες και από άλλα κράτη. Ο κατάλογος ε, που αναφέρεται στο 13β είναι ένας κατάλογος που αφορά άτομα τα οποία έχουν ήδη καταδικαστεί και γι' αυτό λοιπόν θα ήταν σημαντικό εάν ε, στα κράτη-μέλη να μπορεί να αποφασιστεί κατά πόσον είναι δυνατόν να εξάγουν τα άτομα και οντότητες. Θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, ε, όταν εγώ ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών και ασχολιόμουν με θέματα χώρε Βαλτική, τότε μιλάγαμε για τρίτε χώρε. Δεν ήταν χώρε του ΝΑΤΟ, οι χώρε τη ε, Βαλτική. Και τότε έπρεπε να συνυπογράψουμε μαζί με μια άλλη υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι εγκρίνονται ακόμα και οι ε, αμελητές εξαγωγές. Ε, και ξέρετε εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει ήταν ότι όταν πρόκειται να γίνουν εξαγωγές στις αστυνομικές αρχές τότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Αλλά αν κάποιος έμπορος όπλων ήθελε να εξάγει έστω και ένα μικρό πιστόλι ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Τότε βέβαια δεν είχαμε πληροφορίες από άλλα κράτη. Δεν γνωρίζαμε τη δική τους άποψη. Και ως εκ τούτου εκείνος που λάμβανε τις αποφάσεις και αυτός δεν ήταν απαραίτητα πολιτικός, μπορεί να ήταν και σε επίπεδο διοικητικό. Με πάση περιπτώσει, όποιος λαμβάνει τις πληροφορίες ε, θα βοηθούσε πολύ να έχει ενημέρωση για όσους υποβάλλουν έτοιμα που δεν είναι πάντα κράτη, είναι και ιδιώτες έμποροι όπλων που ε, πουλάνε όπλα. Γι' αυτό λοιπόν ε, την αναφορά αυτή στο παράγραφο 13 τη βρίσκω ιδιαίτερα θετική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαφχάουζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, με κύριο Σαφούζερ. Συμφωνώ με κάποιους συναδέρφους. Πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα η επικουρικότητα έχει σαν αποτέλεσμα οι χώρες να έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα. Συμφωνώ με τα κριτήρια. Πιστεύω ότι πράγματι χρειάζεται συντονισμός, αλλά εγώ δεν βλέπω τι παραπάνω έχει να προσφέρει η Ευρώπη και γιατί. Ήτανε κατά η Ευρώπη του πολέμου στο Ιράκ, τότε ήμουν φίλος με τον κύριο Πέτερινγκ που ήταν ε, πρόεδρος ε, της, ε, μάλλον πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ήμασταν κατά. Και ήρθε μετά να με βρει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για να μου μιλήσει εναντίον των αποφάσεων αυτών τα ίδια και μετά Ουκρανία και λοιπά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδειξε να είναι προσεκτική σε όλες αυτές τις ε, υποθέσεις που κατέληξαν σε πόλεμο. Τον πόλεμο πρέπει να τον προλαβαίνουμε και όχι να ασχολούμεθα μόνο με τις συνέπειές του. Και αυτό θα γίνει αν ελέγχουμε τις εξαγωγές όπλων. Υπενθυμίζω ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κοσυφοπαίδιο επίσης οδήγησε σε εξάπλωση όπλων και έλλειψη ελέγχου δεδομένων ε, των ε, θέσεων που πήραν ε, διάφορες χώρες και αυτό το κομμάτι της συγκεκριμένης χώρας. Και εδώ συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν για τη Σαουδική Αραβία. Η χώρα μου πρώτα απ' όλα πρέπει να κατηγορηθεί για ό,τι έκανε. Αλλά αυτό δεν είναι δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι δουλειά του Εθνικού Κοινοβουλίου, τη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Είναι θέμα ελέγχου, αλλά και θέμα συμφερόντων, συγκρούσεων. Πρέπει να καταδικαστεί. Μπορεί να υπάρχει και έγκλημα ε, προδοσίας εδώ και για να επανέλθω στο θέμα μας, να ενισχύσουμε τις εθνικές νομοθεσίες, σίγουρα να φροντίσουμε να έχουμε στη διάθεσή μας κοινά κριτήρια, να στηρίξουμε τα 8 κριτήρια, αυτό πιστεύω ότι είναι καλό, να συντονιστούμε μεταξύ μας, αλλά μην βάζουμε κυρώσεις ή κυδαιμονία μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βαλέρο και πάλι. Παρακαλώ κυρία Βαλέρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, άκουσα προσεκτικά, ε, σημείωσα και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε τελικά πάνω στα διάφορα ζητήματα πριν φτάσω εδώ ήδη ήξερα τι ε, τροπολογίες θα θέλατε να υποβάλλετε γιατί έχουμε συζητήσει για όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά είμαι έτοιμη να συνεχίσω να συζητώ μαζί σας και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Αυτό κάναμε και την προηγούμενη φορά, για την προηγούμενη έκθεση. Αν μάλιστα δεν με απατάει η μνήμη μου, τότε επίσης είχαμε μιλήσει για κυρώσεις που θα έπρεπε να επιβάλλουμε σε όσους δεν τηρούν τα κριτήρια. Ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε λοιπόν και να συμφωνήσουμε για αυτά τα θέματα. Περιμένω τις τροπολογίες σας και για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν τόσο πολύ άριθμοι που πήρατε σήμερα το λόγο και αντιδράσατε στο δικό μου σχέδιο έκθεση. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Συναδελφοί, σας θυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι αύριο μέχρι τις 11 το πρωί, έτσι. Αύριο 11, όχι όπως συνήθως που είναι 12, τώρα είναι 11 το πρωί. Και θα εγκριθεί στην ΑΦΕΤ στην... Μάλλον θα, στις 21-22 Ιουνίου πρώτα θα εγκριθεί στη δικιά μας επιτροπή έκθεση αυτή, μετά στην ΑΦΕΤ 10 ή 11 Ιουλίου. Σωστά. Και στην Ολομέλεια θα πάει για ψηφοφορία το ζήτημα το Σεπτέμβριο, φαντάζομαι, δεν ξέρω πότε ακριβώς. Εντάξει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και για την συζήτηση αυτή που είχαμε. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη τώρα είναι ενημέρωση σχετικά με την αποστολή της ε, ΣΕΝΤΕ στην Κόμα και στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Τρεις βουλευτές, μέλη της ΣΕΝΤΕ, ήταν στην ε, αντιπροσωπή αυτή ο κύριος Χαβιέρ Νάρτ, ο κύριος Σαλίκ ε, Σαφοζέρ και εγώ ίδια που πρίδρευα της αποστολής αυτής. Μας συνόδευσαν και μέλη της Γραμματείας, πολιτικοί σύμβουλοι και βεβαίως και κάποιοι διερμηνείς. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε υποβάλει έκθεση, κάτι γραπτά, οπότε η ενημέρωση θα είναι προφορική. αν χρειαστεί, όταν υποβληθεί το γραπτό κείμενο, θα δούμε αν χρειαστεί να το συστήσουμε και να το εγκρίνουμε. Έτσι κι αλλιώς στην Ολομέλεια έχουμε το θέμα αυτό, την κατάσταση ασφάλειας δηλαδή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θα γίνει συζήτηση, έχουν ήδη υποβληθεί ψηφίσματα Χτες ήταν η λήξη της προθεσμίας, οπότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για την αποστολή αυτή. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ενημερωτική αποστολή. Δεν πήγαμε στην πρωτεύουσα και μετά στην κόμμα από την Αντίσα Μπέμπα πήραμε πτήση κατευθείαν. Οι διευθυντές ήταν πάρα πολύ καλές. Είδαμε πρώτα εκπροσώπους της κυβέρνησης του Κιβού, της επαρχίας του Κιβού και η συνάντηση αυτή καθόλου παρά ικανοποιητική ήταν πρέπει να πω. Μας παρουσιάστηκε μια λαμπρή εικόνα όσον αφορά την πολιτική κατάσταση. με το που φτάσαμε έγιναν διάφορες δηλώσεις από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες δυτικές δημοκρατίες για την ανησυχία τους όσον αφορά την κατάσταση στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Τα κύρια στοιχεία στην ημερήσια διάταξη πάντως ήταν συνάντηση με το Μανούσκο που είναι η αποστολή του ΟΗΕ που βρίσκεται επί εκεί στο ανατολικό τμήμα της χώρας Συναντηθήκαμε επίσης και με άλλες οργανώσεις, την ΟΤΣΑ και την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε με ε, την ηγεσία της περιφέρειας. με το FARDC. Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνάντηση αυτή από την άλλη πλευρά. Τα συμπεράσματά μας από την συνάντηση με το Μανούσκο ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Μάλιστα πριν από εκλογές που πρέπει να λάβουν χώρα εκεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς περιμένουμε. Η διαδικασία καταγραφής των ψηφοφόρων ήταν επιτυχής από ό,τι φαίνεται από τις πρώτες εκτιμήσεις που έχουν γίνει. Το στρατηγείο της Μονούσκο μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν τώρα εμπόδια προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διαδικασία αυτή εγγραφή στους ε, εκλογικού καταλόγους των ε, ψηφοφόρων. Πάνε καλά τα πράγματα σε όλη τη χώρα και βάσει του χρονοδιαγράμματος. Βέβαια, η Δημοκρατία του Κονγκό είναι μια τεράστια χώρα και είναι πολύ δύσκολη η διαχείρισή της. Όμως, ήδη εδώ και χρόνια γίνονται εκλογές σε αυτή τη χώρα και η κατάσταση της ασφάλειας δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ ώστε να αναβληθούν οι εκλογές. Στις συναντήσεις λοιπόν που είχαμε με την ηγεσία της Μονούσκο και με εμπειρογνώμονες οι προβουλευτές μας είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρμογή της τρέχουσας εντολής. Γίνονται έργα για να τροποποιηθεί η εντολή και να μπορέσουν στρατεύματα να εμπλακούν σε περιοχές που υπάρχουν συγκρούσεις τονίσαμε με τους εκπροσώπους του ΟΗΕ την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την εξόρυξη ορυκτών που αποτελεί και μία από τις αιτίες πολλών συγκρούσεων. Και είναι αιτία και γερμανωμένο έγκλημα. Πρόσφατα, λοιπόν, είχαμε δολοφονία εμπειρογνωμόνων του ΟΙΕ υψηλά εστάμενων. που βρίσκονταν εκεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει στείλει ερευνητική αποστολή ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για να διερευνήσει την υπόθεση. Αφού επιστρέψαμε στις Βρυξέλλες αποφασίστηκαν στοχευμένες κυρώσεις κατά του πολιτικού καθεστώτος της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό. Κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά ήταν βάση των όσων περιμένουμε, ήταν αναμενόμενα. Θελήσαμε να πάμε και στο IDP, στο καταβλισμό εκεί, για να συναντηθούμε με εκπροσώπους και με επικεφαλής στον ε, καταβλισμό αυτό που βρίσκονται εσωτερικά εκτοπισμένοι. Μας είπαν ότι αυτός ειδικά ο καταβλισμός της Μουγκούγκα θα διαλυόταν και ότι αυτοί οι εκτοπισμένοι έχουν ήδη πάνω από 10 χρόνια σε αυτόν τον ίδιο καταβλισμό και ότι θα έπαιρναν πια, θα είχαν ένα διαφορετικό καθεστώς μέσα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γκόμα είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος, πολύ κοντά σε ενεργά ηφαίστεια. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένοπλες επιθέσεις, για παραβιάσεις, πρέπει να έχουμε υπόψη μας και την δύσκολη κατάσταση που ζουν οι άνθρωποι αυτοί και αυτοί που έρχονται από άλλες αφρικανικές χώρες ή από άλλες επαρχίες αν τυχόν υπάρξει έκρηξη στο ηφαίστειο που βρίσκεται εκεί πιο κοντά, τι θα γίνει. υπάρχουν ε, και μεγάλα προβλήματα υγείας. Η πρωτεύουσα της επαρχίας βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρουάντα. Και εκεί η πολιτική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και επηρεάζει. Υπάρχουν ε, και ιστορικά γεγονότα που δυσκολεύουν την ε, ασφάλεια στην κάμα. Θα ολοκληρώσω τις παρατηρήσεις μου λοιπόν εδώ για αυτή την επίσκεψη. Και υπόσχομαι ότι όσο γίνεται πιο γρήγορα θα υπάρξει γραπτό κείμενο και θα σας σταλεί. Τώρα, οι άλλοι συμμετέχοντες στην αποστολή, τι έχουν να προσθέσουν. <coughs> Ο κύριος Χαβιέρ ένα κείμενο μπορεί να κρύβει και ψέματα τα οποία διοικητικά φαίνονται αλήθεια. Αυτό εγώ που είδα στην κόμμα πάντως είναι το παράδειγμα της υποκρισίας, του ψέματος όσον αφορά την προσπάθεια ειρήνευσης και αυτό με τα χρήματα άλλων. Η Μονούσκο έχει δώσει 1 δισεκατομμύριο 400 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να προστατεύσει, αλλά είναι μια υποκριτική αποστολή προστασίας, όπου 17.000 στρατιώτες, εξοπλισμένοι μέχρι τα δόντια και με αρκετό υλικό για να επιβάλλουν την ειρήνη, κυκλοφορούν, όπως λένε οι ντόπιοι, σαν τουρίστες στους δρόμους. Η πραγματικότητα είναι ότι παραβιάζουν συστηματικά την εντολή. Η εντολή των Ηνωμένων Εθνών λέει ότι αυτοί οι 17.000 στρατιώτες που τους πληρώνει ο κόσμος ολόκληρος είναι να εξουδετερωθούν οι ένοπλες ε, δυνάμεις εκεί και να προστατευτεί ο πληθυσμός. Αυτή είναι η εντολή που έχει ο ΙΕ. Η εξουδετερώση τέτοιων ένοπλων ομάδων σημαίνει ότι θα έπρεπε Όντω να εξαφανιστούν αυτές οι ανοπλέ ε, ομάδες. Και όταν μίλησα με τον ε, αρμόδιο των ε, δυνάμεων της Μονούσκου από την Νότια Αφρική, μου είπε όντω ότι σημαίνει καταστροφή των ομάδων αυτών. Σημαίνει να σκοτωθούν οι ομάδες αυτές, να φυλακιστούν και να παρετηθούν. Αντιπαράθεση σημαίνει. Είναι ξεκάθαρο. Οι μονάδες της Μονούσκο όμως τι κάνουν. Βρίσκονται έξω-έξω στην αρχή των μεγάλων λιμνών και ειρηνικά κυκλοφορούν στους δρόμους. Οποιοςδήποτε γνωρίζει την περιοχή καταλαβαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, το μεγαλύτερο μέρος ε, των ε, πόρων που δεν είναι τόσο κοβαλτιό, είναι πιο πολύ χρυσός που βρίσκονται όμως ε, αυτοί βρίσκονται μακριά από εκεί που βρίσκονται αυτές οι ένοπλες ομάδες που εκμεταλλεύονται τους πόρους. Πρόκειται για συμμορίες από τον Πακλαντέ, στην Ινδία και αλλού Συγγνώμη, στη, στη Μονόσκου υπάρχουν άνθρωποι από τις χώρες αυτές που τους πληρώνουν ΙΕ και οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο, δεν βρίσκονται εκεί από ιδεολογία, βρίσκονται εκεί γιατί εκεί έχουν βρει δουλειά και εκεί τους πληρώνουν. Και δεν απομακρύνονται από τους κεντρικούς δρόμους για να πάνε να βρούνε και να έρθουν σε αντιπαράθεση με τις ανώπλες ομάδες. Συνεπώς, υπάρχει αυτή η εντολή εξουδετέρωσης των ένοπλων ομάδων και το σκανδαλώδες είναι ότι δεν το κάνουν, δεν κάνουν τίποτα τέτοιο. Όντω πήγαμε στον καταβλισμό της Μουγκούγκα 6-7 χιλιόμετρα από την κόμμα. Εκεί οι γυναίκες μας ζητούσαν κάτι που δεν χρειάζεται μια ειδική αποστολή απλώς να τις προστατεύουμε για να μην κινδυνεύουν από βιασμό όταν πάνε να βρουν νερό. Και όλα αυτά 6 χιλιόμετρα από εκεί που είναι η έδρα της ε, δύναμης αυτής του ΟΗΕ. Μα είναι σκανδαλώδες, είναι αναξιοπρεπές. Δεν μας ζήτησαν τίποτα φοβερό, μόνο αυτό μας ζήτησαν, να τις προστατεύσουμε από το βιασμό. Υπήρξε ψήφισμα, δεν ξέρω από πού, που λέει ότι πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τη δράση της Μανούσκου. Μα εγώ καταργέμαι τη δράση αυτή της Μανούσκου και των γραφειοκρατών του ΟΗΕ. Η Μανούσκου λοιπόν πρέπει πρώτα απ' όλα να ασκεί την εντολή της. Αυτό σημαίνει να πρόκειται για δυνάμεις που θα εκτελέσουν την εντολή τους. Δεν θα κυκλοφορούν σαν τουρίστες. Δεύτερον, αυτός που είναι επικεφαλής τώρα είναι ένας κατάλληλος επικεφαλής, αλλά που δυστυχώς δεν μπορεί να φέρει σε πέρα στην εντολή του, γιατί η εντολή του είναι αυτή που είναι τραυματισμένη. Από τις 17.000 άντε 3.500 να δραστηριοποιούνται πραγματικά, οι υπόλοιποι κάνουν βόλτα. Ενώ η εντολή τους είναι να πάνε σε αντιπαράθεση με τις ένοπλες αυτές ομάδες. Δεν χρειάζονται όλοι αυτοί. Λιγότεροι χρειάζονται. Όταν υπάρχουν 4-5 χιλιάδες ε, από τις διάφορες συμμορίες, δεν μας χρειάζονται 17 χιλιάδες. Χίλιοι, δύο στρατιώτες θα φτάνανε από τη Μονούσκο, αν όντως και πραγματικά βρίσκονταν εκεί για να αντιμετωπίσουν τις ε, συμμορίες. Αλλά δεν το κάνουν. τη δικιά τους τη ζωή προστατεύουν, κανενός άλλου. Και θέλουμε και κάτι άλλο. Η λογιστική του πολέμου, πώς συνδυάζεται με το εμπόριο του χρυσού και άλλων πόρων. Με αυτό ασχολούνται άνθρωποι και από το Κονγκό αλλά και εκτός Κονγκό. Τη Ρουάντα για παράδειγμα. Και υπάρχουν σκοταλόγους του ΙΕ. Τους ξέρουν. Οι υπηρεσίες έρευνας με τις οποίες μίλησα στην κόμμα έχουν 200 θέσει που είναι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι διάφορους ε, πολιτικούς υπεύθυνου που ασχολούνται με αυτό το παράνομο εμπόριο, αλλά δεν υπάρχουν στον κατάλογο για κυρώσει. Αυτός ο κατάλογος κυρώσει πρέπει να φτάσει στους κύριου υπεύθυνου και όχι στους δευτερεύοντες. Αυτό σημαίνει περιουσιακά στοιχεία να μπλοκαριστούν στο εξωτερικό γιατί τελικά το εμπόριο αυτό των φυσικών πόρων της χώρας καταλήγει στις δυτικές τράπεζες. Και οι πόροι αυτοί καταλήγουν σε χώρες κυρίαρχες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι απλώς κλαίμε για τα θύματα και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαφχάουζερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα αυτά που είπε ο συνάδελφος, ο Χαβιέρ Νάρτ. Γιατί πράγματι και εγώ πιστεύω ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να δεσμευτούμε περισσότερο με κινητά τάγματα 3.000-5.000 άνθρωποι το πολύ θα φτάνανε χωρίς πρόβλημα να σταθεροποιήσουν τη χώρα. Αν ήταν αυτό που θέλαμε. Δεν μπορούμε να παίζουμε με εξωτερικές δυνάμεις όπως είναι η Μονούσκο. Χρειάζεται στρατός, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία. Ξέρουν, είναι σε θέση και το κάνουν να παρεμβαίνουν στο εξωτερικό. Θα έπρεπε λοιπόν να ενισχύσουν τον ε, τοπικό εθνικό στρατό. Η λύση στη σύγκρουση αυτή είναι πάνω απ' όλα κινητά τάγματα τα οποία να πλαισιώνονται από εξωτερικές δυνάμεις που ξέρουν να κάνουν πόλεμο και τον κάνουν συχνά στο εξωτερικό και που να παρέμβουν κατευθείαν. Διαπιστώνω, το είπε και ο συνάδελφος, ότι από το σύνολο των καταδικασμένων βάζουμε κάποιους πολιτικούς υπεύθυνους από το Κονγκό, αλλά ξεχνάμε αυτούς που είναι από τη Ρουάντα, την Ουγκάντα, που συνδέονται άμεσα με το λαθρεμπόριο. Και εδώ είμαστε επιλεκτικοί, έχουμε επιλεκτική μνήμη και βλέπουμε τελικά πώς οι αξίες, οι, τα οικονομικά συμφέροντα, η ηθική θα έλεγα, είναι πράγματα που χρησιμοποιούνται μονόπλευρα, όπως μας εφέρει. Και υπενθυμίζω και το πλαίσιο της κατάστασης αυτής και εγώ συμμετείχα πολύ σε αυτή τη χώρα. Είναι μια δράση που ξεκίνησε στην Ουγκάντα με τις Αμερικανικές υπηρεσίες και μετά επεκτάθηκε. Ήταν ε, αυτή η δράση των ε, αντιφρονούντων που ορχιστρώθηκε από το εξωτερικό για να βάλουν το χέρι σε πρώτη ύλη. Είναι γνωστά αυτά διάφοροι σύμβουλοι φίλοι του κύριου Κλίντον πήγαιναν στην περιοχή και υπέγραφαν συμβόλαια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί ότι έτσι είναι. Οπότε οι εξωτερικές δυνάμεις, είτε πρόκειται για την Ρουάντα είτε για την Ουγκάντα, χρησιμοποιήθηκαν από άλλες εξωτερικές δυνάμεις προς το συμφέρον τους. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και έτσι δημιουργήθηκε μια ορχιστρωμένη ανασφάλεια από την οποία αποφελείται το οργανωμένο έγκλημα και τα συμφέροντα κάποιων δυνάμεων. Και έτσι οργανώθηκε η κατάσταση στις μεγάλες λίμνες με πολλές χιλιάδες νεκρούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρεμβαίνουμε τώρα. Και με αυτό τον τρόπο πρέπει να φροντίσουμε να προσαρμόσουμε τις κυρώσεις μας ή τις συστάσεις μας ανάλογα. Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ εδώ τώρα στην δημοκρατική μετάβαση. Έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση ιδιαίτερα υποκριτική. Γιατί αυτή η δημοκρατική μετάβαση. Ο πρόεδρος Καμπίλα, όπως το είπε, ας πούμε ότι θα φύγει. Ελπίζω, όντως, να φύγει. Γιατί πιστεύω ότι είναι αναγκαίο για τη σταθερότητα και για την ειρήνη. Πιστεύω όμως επίσης ότι πρέπει να αφήσουμε το χρόνο για να δημιουργηθεί αυτή η δημοκρατική μετάβαση έτσι ώστε αυτή να είναι πραγματική και να μην προσπαθούμε να στηρίξουμε διάφορους ηγέτες που επίσης έχουν ε, ενορχιστρωθεί απαλού γιατί αυτό θα οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, πολλοί έχουν συμφέρον να συνεχιστεί ο πόλεμο. Οπότε εμεί πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί ώστε να αποφύγουμε πάση θυσία πέρα από την επισημότητα τη μετάβαση, ακόμα και αν είναι απολύτω αναγκαία η μετάβαση και τη στηρίζω απόλυτα, πρέπει να αποφύγουμε τον πόλεμο όμω πρώτα απ' όλα. Βλέπετε, κάποιοι που είναι αναμεμειγμένοι σε σκοτεινές υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το οργανωμένο έγκλημα, αλλά από την άλλη επίσημα είναι οργανωμένοι με κοινωνίες, το καλύτερο για αυτούς είναι να παραμείνουν οι ταραχές και η λαϊκή δημοκρατία του Κογκό να μην γίνει ποτέ κυριαρχοκράτος με δικό του στρατό που να μπορεί να υποστηρίξει τα δικά του συμφέροντα. Και κάποιοι το φροντίζουν αυτό ακόμα και πίσω από τη δημοκρατική μετάβαση, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν να χειραγωγούν τη δημοκρατική διαδικασία. Θυμόσαστε ότι προηγούμενος τι είχε γίνει, πώς δολοφονήθηκε εδώ. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο τίμοι και ειλικρινεί όταν μιλάμε για δημοκρατική μετάβαση, γιατί χρειάζεται χρόνο. Πρέπει να στηρίξουμε επίσης τις εκκλησίες τις δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών, που είναι ειλικρινής. Εκεί πρέπει να στηριχτούμε. Χτες υπήρξε μία διάσκεψη με αντιφρονούντες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κακό. Δεν πήγα, αλλά ο βοηθός μου μου είπε ότι η αντιπολίτευση ήταν ο πιο μετριοπαθής ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει περισσότερα από ό,τι ζητάει η ίδια αντιπολίτευση. Όταν λοιπόν μα λένε η ίδια αντιπολίτευση ότι πρέπει να αποφύγουμε τον πόλεμο και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ε, εμεί να μην ερχόμαστε με, με ακρότητε που είναι και υποκριτικέ και που ξέρουμε από πού ξεκινούν και καταλήξουμε σε αντίθετο αποτέλεσμα. Πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία, το είπα και το ξαναλέω, έχω πάει στη χώρα πολλέ φορέ, να αποφύγουμε τον πόλεμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο κύριος Κάβεντις. Του δίνω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ ειλικρινά τα μέλη της Επιτροπής για την ενημέρωση που μας έκαναν σχετικά με την αποστολή και για τις εντυπώσεις που αποκόμισαν. Επιτρέψτε μου να απαντήσω σε ορισμένα ε, σχόλια. Καταρχάς ε, ήμουν σε θέση να σα ενημερώσω πριν την αποστολή και τότε ήδη είχαμε κάποιες ανησυχίες για την ε, τύχη ορισμένων ατόμων εκπροσώπων από τα Ηνωμένα Έθνη. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους και θέλουμε και εμείς να καταδικάσουμε αυτό το γεγονός και να εκφράσουμε επίσης την επιθυμία μας για μια αντικειμενική και αξιόπιστη έρευνα για το τι συνέβη. Αλλά και για να ερευνηθούν άλλες δολοφονίες και περιστατικά βία στην Κάσα. Κάποια από τα σχόλια που άκουσα θα ήθελα να τα σχολιάσω σχετικά με τη Μονούσκο. Να πω ότι και εγώ συμμερίζομαι ορισμένες ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την εντολή της Μονούσκο και τη δραστηριότητά της εκεί. Είναι σαφές ότι η Μονούσκο έχει διάφορες αρμοδιότητες υπό την εντολή της ε, από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ψήφισμα 4 ε, όχι μόνο δυνατότητα στρατιωτικής επέμβασης, αλλά και καταχώρησης και καταγραφής ε, των ψηφοφόρων σε εκλογές. Και σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας φέτος είναι πιο ε, έντονο σχετικά με την ε, αξιολόγηση των επιδόσεων και τον έλεγχο της δραστηριότητας της Μονούσκο εκεί, έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματική ε, εποπτεία της κατάστασης. Σε γενικές γραμμές Ακούστηκε ότι οι διπλωματικές σχέσεις του Κόγκο με τις γειτονικέ χώρες χρειάζονται ε, εποπτεία και χρειάζεται μια διαδικασία αντικειμενικής παρακολούθησης. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς έχουμε στραφεί σε διάφορες κυβερνητικές οργανώσεις, έχουμε στραφεί στην Αφρικανική Ένωση, θέλουμε στενή συνεργασία μαζί τους, ακριβώς γιατί η κρίση στη δημοκρατία του του Κονγκό θα μπορεί να επιληθεί μόνο με συγκεκριμένε δημοκρατικέ εθνικέ δράσει. Τώρα, ε, ακούστηκαν ορισμένε φωνές για λύσεις, για μέτρα και μπορώ να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το ρηκτά που αποτελούν αιτία συγκρούσεων είμαι ε, και εγώ με το μέρος σας, θέλω να συνεχιστούν οι προσπάθειες αλλά επίσης πρέπει να δούμε και ότι αυτά τα ορυκτά είναι ε, έσοδα, πηγή εσόδων για ε, αυτούς που να αγοράσουν όπλα και για αυτές τις ένοπλες ομάδες που ε, δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Τώρα, όπως γνωρίζετε, έχουμε εγκρίνει μία νέα δέσμη κυρώσεων η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 29 Μαΐου. Σε αυτόν τον κατάλογο κυρώσεων δίδεται έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό γιατί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αποφυγή της βίας είναι για μας εκ των όνουκ άνευ και συνοδεύουν αναπόσπαστα τις εκλογές στη Δημοκρατία του Κονγκό. Όμως ε, δεν θα πρέπει αυτό να αποτρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διευρύνει το πεδίο των ακυρώσεων και να τις ε, εντείνει. Ιδιαίτερα σε όσους εμποδίζουν ε, τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Τώρα, Άκουσα μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπατε για τις ένοπλες δυνάμεις του Κονγκό και λυπούμε που δεν μπορούσατε να συναντηθείτε με την FARDC. Νομίζω πως αυτό θα ήταν σημαντικότατο για το έργο σας, ε, για την ε, αποτελεσματικότητα της ε, Μονούσκο και την δυνατότητα αντιμετώπισης των ένοπλων ομάδων. Πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ Μονούσκο και FARDC και νομίζω πως αυτό είναι και το... πρέπει να είναι και το κύριο μέλημά μας. Τώρα, κατά τα άλλα, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, να πω ότι θα, ε, εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή όλες τις συστάσεις που έχετε κάνει, να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύντομα θα ενημερωθούν γραπτώς και τα υπόλοιπα μέλη, έτσι ώστε να μπορέσουν να σχολιάσουν και να συνεισφέρουν στην ε, συζήτηση. Ήδη έχουν συνεισφέρει γραπτώς τα μέλη της ε, αποστολής που μετέβη στο Κονγκό. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη μέχρι τώρα ανταλλαγή απόψεων. Να κάνω μόνο ένα σχόλιο, επιτρέψτε μου. Να πω λοιπόν ότι συμφωνώ με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για το πόσο σημαντικό είναι να συζητηθούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις και η εξάπλωση της βίας από το ΚΑΣΑ σε άλλες περιοχές. Και σωστά αναφέρατε ότι η εντολή της Μανούσκο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 Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Και εδώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον προσκεκλημένο μας. Τον οποίο θα ε, καλωσορίσουμε σε λίγο μόλις έρθει. It's going to be exchange Πρόκειται λοιπόν για μια ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Πρέσβη Σεράνο, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Το θέμα μας είναι η εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, πολύ επικαιρό θέμα. Τον περιμένουμε λοιπόν. Ambassador Σας καλωσορίζουμε κύριε Πρέσβη στη συνάντησή μας ε, η οποία είναι και ιδιαίτερα επίκαιρη. Εχθές είχαμε τη συνέντευξη τύπου ε, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από κοινού με τον Επιτροπο κύριο Κατάινεν που παρουσίασαν το πακέτο άμυνας μία σειρά εγγράφων τα οποία πρόκειται να συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα δηλαδή είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το να συζητήσουμε τα θέματα αυτά στην Επιτροπή μας. Σήμερα, έτσι μας είπαν, θα έχουμε μία κοινή συνέντευξη τύπου της ε, κυρία Μογκερίνη και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Στόλτενμπερκ. Και στη συνέντευξη αυτή, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν τα 42 μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε και να υλοποιηθεί αυτή η κοινή δήλωση ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ που υπογράφηκε πέρυσι στη Βαρσοβία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να μας ε, παρουσιάσετε την άποψή σας και ελπίζω μετά να ακολουθήσει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα το γεγονός ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ και μου δίνει τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ε, στην συνολική στρατηγική για θέματα άμυνας κυρίως. Ε, και όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε κυρία Πρόεδρε, έχουν ληφθεί πολύ σημαντικές αποφάσεις. Αυτές τις μέρες, εχθές, ε, το πακέτο μέτρων για την άμυνα, ένα έγγραφο στοχασμού και συλλογισμού, σχέδιο κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Άμυνας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί ανοίγει η πόρτα για να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας το οποίο θα είναι και καθοριστική σημασία για να αποκτήσουμε νέες δυνατότητες. Και σήμερα στο Συμβούλιο πρόκειται να εγκριθεί μια απόφαση ότι θα μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες ε, για θέματα επιτελείου στον ε, επικεφαλής ε, ο οποίος ε, προείσταται του στρατιωτικού προσωπικού, μια αρκετά μεγάλη σειρά αποφάσεων που ελήφθησαν αυτές τις μέρες. Και βέβαια είχαν προηγηθεί άλλες αποφάσεις που ελήφθησαν από το Συμβούλιο το Μάιο και σημειώθηκε πρόοδος σε θέματα άμυνας. Νομίζω καλά τα πάμε. Με καλό ρυθμό. Ο βασικός στόχος αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε στην άμυνα, ο βασικός αυτός στόχος είναι διτός. Αφενός υπάρχει ένας ε, κύριος στόχος που είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις ε, αμυντικές τους ε, δυνατότητες και επ' αυτού έχουν αναλυφθεί αρκετές πρωτοβουλίες. Νομίζω η σημαντικότερη είναι η εργασία για το «Premium Structure Cooperation και για το Ταμείο Άμυνα στο οποίο αναφέρθηκα, πρωτοβουλίε που δεν συνδέονται επίσημα μεταξύ τους, όμως ε, η μία στηρίζει την άλλη. Αποτελούν λοιπόν ε, καθοριστική σημασία κλειδί για την βελτίωση των αμυντικών δυνατήτων. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι να βελτιώσουμε τα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, διαχείριση κρίσεων θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στις δυνατότητες ε, του στρατιωτικού σχεδιασμού εδώ, σε αυτό το θέμα, υπάρχει και ένας ε, συντονιστικός ε, φορέας με το, που συνδέεται με το CPPC, που είναι το αστικό, το πολιτικό κομμάτι. Ταχεία αντίδραση. Εδώ γίνεται πολύ καλή δουλειά για τις battle groups, τις περίφημες. Επίσης, παρότι πρόκειται για αστικές ή πολιτικές δυνατότητες, αυτό που ενδιαφέρει είναι να αναθεωρήσουμε και το είδος προσωπικού που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, να αναθεωρήσουμε, αν θέλετε, τις προτεραιότητές μας. Και ένα άλλο στοιχείο είναι να συνεργαστούμε και με άλλες πολυμερείς δυνάμεις, η Eurocore, μεταξύ άλλων, να βελτιώσουμε τη συνειδητοποίηση, την ευαισθητοποίηση μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από ε, την βελτίωση της ε, στρατιωτικής ικανότητας και του στρατιωτικού προσωπικού. Και όλα αυτά μέσα από συνεργασία με εταίρους, αυτός είναι ο τρίτος βραχίωνας, αναφερθήκατε στη δουλειά που κάνουμε με τον ΝΑΤΟ. Η δουλειά που γίνεται για την εφαρμογή των 42 προτάσεων. Σύντομα θα έχουμε μία έκθεση που θα παρουσιάσουν η κυρία Μογκερίνη και ο κύριος Στόλτεμπερκ. Αυτά θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο και μετά βεβαίως θα συνεργαστούμε και με άλλους ε, όπως είναι τα Ηνωμένα Αυτή είναι η δομή αυτών που προσπαθούμε να επιτύχουμε και αν το βρίσκεται χρήσιμο ευχαριστώ να μπω και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ ε, θα ήθελα να επισημάνω την ε, συνεργασία με μόνιμες δομές που έχει δύο στόχους, δηλαδή την βελτίωση των στρατιωτικών, της στρατιωτικής ικανότητας και την ανάπτυξη ικανοτήτων που μπορούν να υποβληθούν από τα κράτη-μέλη για να υπάρχει βελτίωση της ικανότητας γενικότερα της στρατιωτικής ε, τις ε, ικανότητες επίπεδο κεντρικό, ακόμα και τις ικανότητες των battle groups. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί στόχοι. Αυτά όλα να γίνουν μέσα από τη συνεργασία. Γιατί κατ' ουσίαν αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι να υπάρχει η καλύτερη συνεργασία των κρατών μελών στην παραγωγή, στην αμυντική παραγωγή, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο υγιή αμυντική βιομηχανία και να είμαστε και η αιχμή του τώρα σε τεχνολογικό επίπεδο. Μας ενδιαφέρει να υπάρχουν κοινέ δράσεις και αυτό σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει και επίπεδο κοινή ε, ικανότητα, Η ΠΕΣΚΟ είναι ένα στοιχείο που μας τα επιτρέπει όλα αυτά. Ε, αναφέρεται στο 42.6 της συνθήκης ε, πρωτόκολλο 10 Εκεί λοιπόν γίνεται λόγος για υποχρώσεις, δεσμευτικές υποχρώσεις μεταξύ των κρατών μελών ακριβώς για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε από κοινού τις ικανότητες ή να υπάρχουν ικανότητες έτοιμες να αναπτυχθούν. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τα κράτη-μέλη οι πρωτοβουλίες των κρατών μελών ε, γίνονται μέσα από ενημέρωση από τα κρατημέλη κατόπιν ακολουθεί ε, απόφαση του Συμβουλίου. Νομίζω τα γνωρίζετε όλα αυτά. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το επίπεδο των ε, φιλοδοξιών, των στόχων και η δυνατότητα μη εξαιρέσεων, μη εφαρμογής εξαιρέσεων. Τα κράτη-μέλη επιθυμούν να υπάρχει ένα άνοιγμα προφανώς ε, πρέπει τα κρατημέλη να αναλάβουν δεσμεύσεις για μεγαλύτερες επενδύσεις ε, στον τομέα της ε, άμυνας, βεβαίως να αυξηθούν οι δαπάνες προφανώς, όμως αυτό που ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και να μην είναι μια κλειστή λέσχη. Τώρα υπάρχουν κάποια άλλα κρατημέλη που λένε όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ΠΕΣΚΟ τα, κάνει, τα καταφέρνει καλύτερα ε, στο να δεσμεύει περισσότερους πόρους και κονδύλια. Μία ισορροπία λοιπόν ανάμεσα στους στόχους και κάτι που να είναι πιο ανοιχτό προς τους άλλους. Ένας από τους τρόπους που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη εξίσωση είναι μέσα από το σύστημα διαχείρισης της ΠΕΣΚΟ. Αυτή τη στιγμή η πρόταση που σας παρουσιάζω είναι που ακριβώς βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Η ε, πρόταση είναι ε, σύστημα διαχείρισης σε δύο επίπεδα όπου όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να συμμετέχουν, να είναι παρόντα σε στο πρώτο επίπεδο της ε, διαχείρισης ψηφίζουν μόνο τα κράτη της ΠΕΣΚΟ, αλλά μπορούν να είναι παρόντα και τα άλλα κράτη ως παρατηρητές. Και υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο που περιορίζεται στα μεμονωμένα προγράμματα που θα ενσωματώσει η ΠΕΣΚΟ. Γιατί στη τελική ανάλυση ε, θα υπάρχουν δεσμεύσει για όλα τα κράτη-μέλη, ε, άρθρο 2 του πρωτοκόλου 10. Και υπάρχουν και ε, σχέδια, προγράμματα, γιατί οι δεσμεύσεις πρέπει να ε, μετατραπούν σε προγράμματα τα οποία ε, θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν μια κοινή ικανότητα. Τέλος, κάθε πρόγραμμα έχει τη δική του την ιδιομορφία και μόνο τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και στις συζητήσεις. Αυτό λοιπόν είναι από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουμε. Οργανώσαμε μια σειρά εργαστηρίων και θα έχουμε άλλο ένα workshop στις αρχές Ιουλίου. Είναι δύσκολο βέβαια να ορίσουμε χρονοδιάγραμμα για το πόσο γρήγορα θα προσπαθήσουμε και πάλι είναι με διαδικασία που ξεκινάει από τα κράτη-μέλη παρότι τη στηρίζουμε και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζουμε και τις δικές μας απόψεις αλλά προσπαθούμε να προχωρήσουμε ε, κυρίως ε, στη φάση της ε, κοινοποίησης η οποία θα είναι κατά το τέλος του έτους. Αλλά και πάλι σας λέω, η απόφαση θα ληφθεί από τα κράτη-μέλη. Εκείνο που επίσης προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι τα προγράμματα, τα οποία γίνονται προγράμματα της ΠΕΣΚΟ, αυτά να χρηματοδοτούνται ε, μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, ε, το οποίο πρόκειται να συσταθεί, θα υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να φέρω είναι η ετήσια αναθεώρηση και αναφορά για θέματα άμυνας. Επ' αυτού ε, λήψαν αποφάσεις το Μάιο και συμφωνήθηκε να υπάρξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη. Αφορά τα κρατημέλη, την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κρατημέλη ε, για ε, εθνικά προγράμματα άμυνας. Τι πρέπει να γίνει για να καλυφθούν κενά. Όπως ξέρετε υπάρχει ένα πρόγραμμα βελτίωση των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνδέεται με τους στόχους μας, τώρα να θεωρείται, αλλά είναι σημαντικό ε, τα κράτη-μέλη να ανοιχτούν, να υπάρχει διαφάνεια ε, στον ε, εθνικό τους αμυντικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς κοινούς στόχους και να μπορέσουμε να καλύψουμε ενδεχόμενα κενά στην ε, βελτίωση των αμυντικών ικανοτήτων. Όλα αυτά ε, συμπληρώνονται από το αμυντικό πρόγραμμα δράσης. Ε, η Κομισιόν έχει καταθέσει μια πολύ φιλόδοξη πρόταση. Το ποσό της και η μορφή της χρηματοδότησης θα κρυφτεί από τη συμφωνία. Το Κοινοβούλιο, ως αρμόδιο για τα δημοσιονομικά, θα έχει εδώ λόγο. 500 εκατομμύρια το χρόνο για την έρευνα, για την επόμενη, προβλέπονται για την επόμενη δημοσιονομική προσεπτική και επίσης και βελτίωση των ικανοτήτων ε, και γι' αυτό προβλέπονται περίπου 500 εκατομμύρια σε ετήσια βάση. Και κατόπιν υπάρχει ενδεχομένως και η δυνατότητα, αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν, να υπάρχουν ε, χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα είναι πέρα από αυτά που προαναφέρθηκαν από την πρώτη φάση. Αυτά όμως εκτός προϋπολογισμού και εδώ υπάρχουν περιορισμοί στο 41-2. Αυτές είναι οι προσπάθειες ε, που ε, καταβάλουμε έτσι ώστε να βελτιωθεί η στρατιωτική ικανότητα της, ε, των κρατών μελών. Όσον αφορά τώρα τη δική μας τη δομή, το πρώτο που πρέπει να επισημάνω είναι η στρατιωτική ικανότητα. Όπως είπα ήδη στην αρχή, τώρα πλέον υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή, έχει αναλάβει αρμοδιότητες, έχει τρεις ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις, αυτές καλύπτει από τις πέντε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι δύο είναι στην Κεντρική Μεσόγειο και οι άλλοι ε, στην ακτή της Σομαλίας και άλλες τρεις είναι κυρίως σε επίπεδο εξάσκησης. Αυτές είναι στο Μαλί, στη Σομαλία. Βλέπετε ότι είναι πολύ δύσκολο το περιβάλλον στο οποίο κινούνται αυτές οι δύο τουλάχιστον τελευταίες, άρα δηλαδή χρειάζονται την υποστήριξη από τα κεντρικά μας από την έδρα μας έτσι ώστε να στηριχτεί ο δικητής ε, που βρίσκεται επιτόπου ε, να μην αναγκασμένος να ασχολείται με γραφειοκρατικά θέματα τα οποία διεκπαιρεώνονται στις Βρυξέλλες. Είναι σημαντικό να προσφέρεται υποστήριξη στον επιτόπου διοικητή ε, κυρίως όταν υπάρχουν κρίσιμες περίοδοι που υπάρχουν τέτοιου είδους περίοδοι στις χώρες αυτές. Αυτά εξελίσσονται από το στρατιωτικό προσωπικό. Ε, θα προσλάβουμε άλλους 20 έκτακτους. Αυτοί όμως ε, θα ενταχθούν γενικότερα στη στρατιωτική δομή, ανταλλαγή πληροφοριών, επιμελητία. Ε, δηλαδή, ίσως αυτά να μοιάζουν αρκετά και δεν υπάρχει ανάγκη για επιπρόσθετο προσωπικό. Η NBCC στηρίζεται από μια, ένα κοινό, μια άλλη κοινή δομή προσωπικό από MPCC και από CPCC έτσι ώστε να υπάρχει συνέργεια στο σχεδιασμό, ε, στην ε, εξέλιξη των επιχειρήσεων. Αυτό, ας πούμε, θα μας επιτρέψει το Μαλί όπου έχουμε και στρατιωτική και πολιτική επιχείρηση, εκεί θα μπορούσαν να μοιραστούν τα κτίρια, ε, την επικοινωνία, την προστασία των ε, δυνάμεων, να υπάρχει καλύτερος ε, συντονισμός της εντολής και όλα αυτά θα μπορούσαν να στηριχθούν μέσα από μια κοινή δομή. Για την MPCC υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρηση για το 2018. Όσον αφορά τα περίφημα battle groups, αυτά είναι ένα σημαντικό θέμα. Αυτά είναι η ε, ταχύ ανάπτυξη ομάδας κρούσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι 2.700 άνδρες καλύπτουμε. 10 μέρες. Μετά από 10 μέρες θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί εφόσον έχει ληφθεί απόφαση. Αυτά για τα battle groups. Και ε, είναι αυτάρκης οι ομάδες αυτές. Πρέπει να είναι αυτάρκης. Νομίζω αυτές συστήθηκαν το 4, το 2004. Ε, η συλλήφθηκε ιδέα, αλλά ποτέ δεν είχαμε αναπτύξει ένα battle group. Είχαν κάποιο σημαντικό ρόλο στο να αλλάξουν οι εθνικές δυνάμεις. Έπρεπε να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να υπάρχουν και δυνάμεις που να αναπτύσσονται σε επιχειρήσεις. Χρήσιμο αυτό για να συνεργαστούν τα κρατημέλη. Ποτέ όμως δεν υπήρξε πραγματικά ανάπτυξη αυτής της battle group. Τα Ηνωμένα Έθνη επιτιμούν διακαώς να υπάρχουν όμως αυτές οι battle groups ε, διότι ε, μπορούν να βοηθήσουν τα μάλα σε πολλές επιχειρήσεις. Τους τελευταίους μήνες εξετάζουμε το ποια είναι τα βασικά εμπόδια για την ανάπτυξη των ομάδων αυτών. Δύο εντοπίσαμε. Η μία είναι, δυσκολία είναι στη χρηματοδότηση. Το να οριστεί κοινό κόστος. Όπως ξέρετε, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ε, χρηματοδοτούνται άμεσα από τα κράτη-μέλη μέσα από το μηχανισμό Αθήνα. Και δεν υπάρχει γενοδορία όσον αφορά τον ορισμό του της ανάληψης, κοινή ανάληψης του κόστους, ε, το οποίο μέχρι τώρα ήταν το 10% του συνολικού κόστους που προκύπτει από μια επιχείρηση. Οι μάχη μέσα αυτές τις ομάδες, οι battle groups, είναι πολύ δαπανηρές, γιατί αναπτύσσονται ε, άνδρες και γυναίκες βέβαια, στρατιώτε, ε, με εξοπλισμό σε σύντομο χρονικό διάστημα, άρα κόστο μεταφορά. Όλα αυτά είναι πολύ δαπανηρά και υπήρξε ήδη μία δήλωση η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο ε, θα καλύπτεται η ανάπτυξη. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα, μεταφορά, επικοινωνίες, ε, επιμελητεία. Αυτά δεν καλύπτονται, δεν είναι κοινά αναλαμβανόμενο κόστος από όλους δηλαδή. Το Μάιο οι Υπουργοί συμφώνησαν να εξετάσουν αρκετά θέματα, ανάπτυξη, ξανά ανάπτυξη, βασικά στοιχεία υποστήριξης, για να διαπιστωθεί κατά πόσον με αναθεώρηση του μηχανισμού Αθήνα, ε, που υπάρχει έτσι κι άλλως αυτή τη στιγμή, να δουν λοιπόν ε, κατά πόσον μπορούν να συμπεριληφθούν σε κοινή ανάληψη κόστους ε, περισσότερα στοιχεία. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τα battle groups, δεν υπάρχει standard, δεν υπάρχουν μόνιμες τέτοιες ομάδες, που σημαίνει κάθε φορά και κάθε ομάδα ε, συστήνεται με διαφορετικό τρόπο. Μερικές ενδεχομένως είναι καλύτερες για ε, θαλάσσιες επιχειρήσεις, άλλες πάλι για άλλες μορφές επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου ε, πρέπει να υπάρχουν κάποια μοντούλα, αν θέλετε, που να μπορούν να ταιριάζουν ε, σε κάθε battle group που συστήνεται, να υπάρχουν ε, διάφορες δυνατότητες έτσι ώστε να προσαρμόζεται η ομάδα. Και αυτά μπορούν να γίνουν μέσα από την ΠΕΣΚΟ. Άρα αυτή είναι μία από τις χρησιμότητες της ΠΕΣΚΟ. Αυτό είναι το Battle Group Plus και υπάρχει και Battle Group μείον. Δηλαδή σε ορισμένε περιπτώσει πρέπει να υπάρχει ταχύτατη ανάπτυξη, αλλά όχι του συνόλου του battle group, μόνο ορισμένων στοιχείων της ομάδας. Και εδώ ορισμένα κρατημέλη είναι επιφυλακτικά, ε, δεν το επιθυμούν ε, πολύ. Ε, υπάρχει αυτό, υπάρχουν και δύο battle group ε, ε, όπου είναι σε αναμονή ανά Πολλοί λένε ότι αυτό δεν είναι καλή χρήση των ομάδων αυτών. Εγώ πιστεύω ότι καλύτερα να ε, αναπτύσσονται οι ομάδες ε, παρά να βρίσκονται εν αναμονή. Με πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση γιατί πιστεύω ότι αυτό θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά μας. Έχω μιλήσει πάρα πολύ. Tell me when to stop. Uh, but maybe just to mention also civilian capability. Κάτι άλλο, ναι, είναι η ανάπτυξη, η ικανότητα ανάπτυξη των πολιτών για θέματα άμυνας. Όμως, όπως γνωρίζουμε, η ασφάλεια και η άμυνα είναι μια ευρύτερη έννοια και φυσικά οι ικανότητε των πολιτών έχουν αποδειχθεί πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αναπτύξουμε μηχανισμούς για να αυξηθεί η ταχύτητα ανταπόκριση, είτε εδώ στο κεντρικά είτε σε μέρη που έχουμε εντοπίσει όπου υπάρχει ανάγκη γι' αυτό και σε στάδιο του σχεδιασμού και ε, με την παρουσία μας εκεί και τη βοήθεια στις νομικές αρχές. Συνεχίζεται λοιπόν η δουλειά εκεί για να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι μηχανισμοί που θα μας επιτρέψουν να το πράξουμε και μετά εξετάζουμε την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων. Ε, αναφέρθηκα στις ικανότητες των πολιτών ήδη. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τομείς ε, που ισχύουν από το 2000 ε, διοίκηση, πολίτες, πολιτική προστασία και αστυνομία. Και αυτό θα βοηθήσει να δημιουργηθούν οι ικανότητες ανάπτυξης που αναφέραμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Και 16 χρόνια μετά τα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι θέλουν να δουν αλλιώς τα πράγματα. Υπάρχει μια αρκετά κάθετη προσέγγιση, βασισμένη σε κατηγορίες και το σκεπτικό τώρα είναι να αλλάξει αυτό και να γίνει μια οριζόντια προσέγγιση, να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε και τι χρειαζόμαστε από πλευρά προσωπικού για να το πετύχουμε. Τώρα, θέματα προσωπικού. Ε, σε ό,τι αφορά τις ε, ικανότητες που αναπτύξουν οι πολίτες, εννοούμε τους επαγγελματίες που θα παντρώσουν τις αποστολές. Για επαγγελματικέ ικανότητες, όταν γίνεται λόγος, εννοούμε ε, το hardware, το υλικό, το τεχνικό που θα χρειαστεί. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς από την άμυνα, από τις μηχανές θα περάσουμε στους ανθρώπους, ε, στους πολίτες. Και φυσικά βέβαια ξέρω πως αυτή η σύγκριση δεν είναι δικαίη διότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα σημαντικότερος. Αυτά για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ενημερωθείτε για την πρόοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ωραία. Όπως σας είπα και στην αρχή, είπα ότι εκπρόσωπος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα θα παρουσιάσουν μια κοινή έκθεση, μία, κοινική για τους δύο οργανισμούς, η οποία θα παρουσιαστεί επίσημα και θα δημοσιευθεί εν μέρη στο επόμενο Συμβουλίο, νομίζω στις 19 Ιουνίου. Η έκθεση αυτή θα εξετάζει τις 42 ομάδες κοινών δράσεων, θα εξετάσει σε ποιο στάδιο εφαρμογή είναι. Έχουν γίνει πάρα πολλά μέχρι τώρα, πρέπει να πω, και σε επιχειρησιακές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μεσόγειο, όπου υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία ακτοφυλακής και ε, των μελών της επιχείρησης Σοφία. Επίσης, τα υβρίδια είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Υπάρχουν οι σχετικές 10 ε, ομάδες δράσεων και τα σχετικά έγγραφα. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε ένα, ένα υβρίδιο έτσι ώστε να μπορούμε στο μέλλον να ε, διαχειριζόμαστε από κοινού τέτοια θέματα. Και μετά βρίσκεται υπό επεξεργασία η στρατηγική επικοινωνίας. Μετά, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και ενισχυμένη συνεργασία ε, στα διάφορα θέματα κυβέρνο χώρου. Μετά να πω επίσης, ξέχασα πιο πριν, ότι με τη Φιλανδία είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία σε ό,τι αφορά τα υβριδικά μας ε, παρήχαν εμπειρογνώμονες και εμπειρογνωμοσύνη. Τώρα, αυτή, αυτό τον καιρό τρέχει μία παράλληλη συντονισμένη άσκηση μαζί με το ΝΑΤΟ. Φέτος ε, ηγείται το ΝΑΤΟ της άσκησης αυτής. Και εδώ υπάρχει ένα υβριδικό σενάριο και την ε, εβδομάδα πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, αρχίσει τη δράση η οποία μετά θα συμπεριληφθεί στην ε, άσκηση του ΝΑΤΟ. Το μήνυμα που προσπαθούμε να στείλουμε είναι ότι συνεργαζόμαστε, ότι αντιμετωπίζουμε από κοινού την υβριδική αυτή πρόκληση και νομίζω πως έτσι θα στείλουμε και ένα πολύ δυνατό πολιτικό μήνυμα. Τώρα, βιομηχανική ανάπτυξη, ανάπτυξη ικανοτήτων και αυτό είναι προς όφελος της συνεργασίας μας, προς όφελος του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές εντοπισμού των αναγκών μέσα στα πλαίσια του σχεδίου αυτού. Το σχέδιο, όπως σας είπα, είναι κοινό και υπάρχουν ανταλλαγές απόψεων ε, στις ομάδες μας έτσι ώστε να αποφευθούν υπερκαλύψεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ήδη έχει επαναλάβει πόσο σημαντικό είναι να είναι κοινέ οι προσπάθειες έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές. Νομίζω πως τώρα έχω καλύψει τα περισσότερα θέματα, ξέχασα τους εταίρους. Ναι, ε, αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ και στο θέμα των εταίρων. Έχουμε εντοπίσει τρεις χώρες οι οποίες ε, είναι ενδιαφέρουσες για να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα project, Αζερβαϊτζάν, Μολδαβία, εκείνη την περιοχή. Μετά είπα ότι εκπρόσωπο, επιμένει να δούμε τι έχει αλλάξει σε αυτές τις 42 κοινέ ε, ομάδες δράσεων. Και αυτό που έχει αλλάξει νομίζω πως μπορεί να συνοψιστεί στο εξή το πώς συνεργαζόμαστε. Η συνεργασία πλέον έχει γίνει το σύνηθες, ε, συναντιόμαστε Τακτικά κάθε εβδομάδα εξετάζουμε από κοινού τις προκλήσεις μας και τον τρόπο αντιμετώπισης. Αυτό λοιπόν έχει γίνει τον τελευταίο καιρό. Έτσι προχωράει η συνεργασία μας με τον ΝΑΤΟ και νομίζω πως ήδη μίλησα για πολλή ώρα, οπότε θα σταματήσω εδώ και θα σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να τοποθετηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ και πρέσβη. Σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ η ενημέρωση που μας κάνατε για τα γεγονότα που θα προηγηθούν του Συμβουλίου. Τώρα θα δώσω το λόγο σε εσά. Ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιάστηκα, ομολογώ, και είμαι πολύ χαρούμενος και ταυτόχρονα ευγνώμων για αυτά που άκουσα από εσάς σήμερα, για αυτά που δημοσιεύτηκαν επίσημα χθες. Γι' αυτό λοιπόν και τα καλωσορίζω θερμότατα. Είναι, πιστεύω, ε, αυτά που εμείς ζητούσαμε εδώ και χρόνια. Είναι η προοπτική που είχαμε για το μέλλον, ιδιαίτερα η θέση του ΕΛΚ Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως ε, αρχικά μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένος για το ότι έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια, στα ψηλά γράμματα. Και εδώ αναφέρομαι στα εξή, θα μιλήσω επιγραμματικά. Ε, συμφωνώ σε γενικέ γραμμέ με αυτά που είπατε για τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζω και τι τρει χώρε εταίρου που μα είπατε πώ εντοπίσατε. Ε, η Βοσνία, μία από αυτές τις ε, τρίτες χώρες, είναι μία χώρα που έχει διαφοροποιηθεί ανάμεσα σε σχέση με τις υπόλοιπες της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Τώρα, Μολδαβία, Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ανάμεσα στον πρόεδρο και την ε, κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας. Την Ισία υπάρχει μια γενικότερη πολιτική συνένεση και θα ήθελα να πω επίσης ότι Συμφωνώ απόλυτα για αυτά που είπατε με, σχετικά με τη χρηματοδότηση του μηχανισμού Αθηνά. Νομίζω πως επιτέλους έχει έρθει η ώρα να υπάρξει μια διεύρυνση του πεδίου, όπως είπατε κι εσείς. Γι' αυτό και ήμουν μέχρι τώρα κάπως διστακτικός. Ναι, δεν υπάρχουν οι, δυνα... οι όμως χρειάζονται χρηματοδότηση για περαιτέρω επέκτασή τους. Γι' αυτό λοιπόν ε, χρειάζεται προσοχή σε αυτό διότι υπάρχει μεν η δυνατότητα, αλλά δεν υπάρχουν τα κονδύλια. Τώρα, ε, το Συμβούλιο επιτέλους ε, αποφάσισε το τι θα πράξει στη συνέχεια, αλλά έχω μία ερώτηση. Ποια είναι η λογική ακολουθία εδώ, τι θα γίνει στη συνέχεια. NPCC για τις μη εκτελεστικές αποστολές. Το λογικό θα ήταν να λέμε στο μέλλον ότι εντάξει, το εκτελεστικό σκέλος των αποστολών θα τον αλάβουμε εμείς. Αλλά ε, η CPCC, οι πολίτες που τοποθετούνται σε σχέση με τις στρατιωτικές ε, αποστολές, με τις NPCC. Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, τη θέση αυτή και να καθορίσουμε για τους στόχους σε σχέση με με το ΠΕΣΚΟ. Πρέπει να δούμε ότι δεν έχει αναφερθεί το inclusiveness, όπως το λέτε, ως το ύψιστο επίπεδο των φιλοδοξιών μας. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ε, πιο περιεκτική. Πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές και αυτό πρέπει να διακρίνει την στρατηγική μας ως τα υψηλότερα επίπεδα. Μην ξεχνάτε ότι τα αρχικά PESCO σημαίνουν Permanent Structure Cooperation. Συνε... μόνιμη συνεργασία για τις δομές και όχι συντονισμός και όχι coordination. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω οι φιλοδοξίες μας να είναι ε, τόσο υψηλές που θα ξεπεράσουν τα επίπεδα ΠΕΠΚΟ. Ακούσαμε και για τα κοινά project τα οποία θα χρηματοδοτηθούν, θα συγχρηματοδοτηθούν από το Κοινοταμείο Ασφάλειας. Σίγουρα τα κάτι μέλη θα συνεισφέρουν ε, το μεγαλύτερο ποσοστό των ε, κονδυλίων που ε, χρειάζονται, αλλά θα μπορούσαμε και να προσθέσουμε ένα 10-15% ε, στα κονδύλια αυτά από το πρόγραμμα Juncker. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα ξεκάθαρα λόγια σας, για την ανάπτυξη ικανοτήτων ότι πρέπει να φτάσουμε σε, ένα, σε δημιουργία πρωτοτύπου και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω εάν μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε σε ό,τι αφορά το, σχέ, το σχέδιο νόμου για την αμυντική βιομηχανία, εάν έχουμε επιτέλους τους πρώτους κανόνες για το τι θα γίνει μετά το Brexit για το ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό το project, ε, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν θα είναι όλα οι συμμετέχοντες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς και το Συμβούλιο να έχουμε μία πρώτη εικόνα του τι θα γίνει μετά τον Brexit και τι θα απογίνουν και οι Βρετανικές επιχειρήσεις οι οποίες πλέον θα μείνουν εκτός. Αυτά από μένα προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ και αναμένω με ανυπομονησία την εφαρμογή των, όλων, των όσων μας είπατε. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πάσκου. Με τη σειρά μου θα εκφράσω την ίδια ικανοποίηση και αυτό για το ότι όσα εδώ μας παρουσιάσατε αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται, να λαμβάνεται δράση και είναι αλήθεια ότι τα τελευταία δύο χρόνια κάναμε περισσότερα από ό,τι είχαμε κάνει τα τελευταία 58 χρόνια για αυτό το θέμα. Και όλοι βέβαια το ίδιο ακριβώς ζητάμε από το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να, τώρα το έχουμε. Όμως θέλω να έρθω σε κάποια κάπως πιο συγκεκριμένα προβλήματα και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν τόσο λεπτομερείς για όλα αυτά τα προγράμματα και τα σχέδια. Η κατάσταση τώρα με την ΠΕΣΚΟ και τα σχέδια, και εδώ έρχομαι σε αυτό που είπε και ο κύριος Γκάλερ, η ΠΕΣΚΟ θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από σχέδια και προγράμματα. Πάντως, στο στάδιο που βρισκόμαστε, θυμάμαι την κατάσταση που είχαμε στο ΝΑΤΟ με τη δεκαετία του 90, μετά την εταιρική σχέση για την ειρήνη. Για αυτούς που συμμετείχαν ενεργά και που μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο άρθρο 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, που τότε ήταν η μόνη ε, διασφάλιση και εγγύηση για ασφάλεια που υπήρχε τότε. Οπότε, εγώ ρωτάω, πόσες ασκήσεις έχουμε για να συμμετέχουμε ώστε να θεωρηθούμε ενεργοί συμμετέχοντες και να μπορούμε να αποφεληθούμε από το 4. Αν κάποιος συμμετέχει σε ένα σχέδιο στην ΠΕΣΚΟ, έχει δικαίωμα ψήφου. Είναι η ίδια ιστορία δηλαδή που είχαμε τότε που επανέρχεται μετά από 20 χρόνια. Δεύτερον, οι battle groups, οι ομάδες μάχης. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι καλό που δεν έχουμε ένα μοντέλο, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές καταστάσεις όπου μπορεί να ζητηθεί στο μέλλον να στείλουμε τέτοιες ομάδες μάχης. Και αν έχουμε ένα μόνο μοντέλο, δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση που θα υπάρχει επί τόπου υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές και είναι καλό αυτό. Συγχρόνως είπατε ότι αυτές οι διαφορές μπορούν να επιτρέψουν και περισσότερες ανταλλαγές. Αλλά ωραία, ας πούμε ότι έχω μια κατάσταση όπου χρειάζομαι κάποια στοιχεία που ανήκουν σε μια άλλη ομάδα μάχης. Έχω δημιουργήσει μια ομάδα μάχης για αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά έτσι αφαιρώ στοιχεία από την άλλη ομάδα μάχης. Έτσι θα είναι ή δεν θα επηρεάζονται οι άλλες μάχες ομάδες. Ομάδες μάχης, Διότι δεν θα πρέπει να αποζημούμε τις άλλες ομάδες μάχης για να εξοπλίσουμε τη δικιά μας, την καινούρια. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και το τελευταίο, το ΝΑΤΟ μετά το 2000 πέρασε από την εδαφικότητα στην έννοια περισσότερο της αποστολής. Αυτή η εδαφική άμυνα δηλαδή τέλειωσε. Τώρα έχουμε μόνο δυνάμεις βάσει αποστολών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τώρα πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και συγχρόνως πρέπει να παραδεχτώ ότι η εδαφική μας άμυνα, γενικά μιλώντας, στηρίζεται από άλλα στοιχεία, από άλλους παράγοντες που διαθέτουμε. Αυτά ήταν ένας προβληματισμός από τη δικιά μου την πλευρά, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Η κυρία Λέζινγκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ για την περιεκτικότατη παρουσίασή σας. Οι ερωτήσεις μου αφορούν κυρίως ε, κάποιες ε, λεπτομέρειες που δεν άκουσα σχετικά με τους στόχους ε, του σχεδίου εφαρμογής. Νομίζω πως είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Έχει ζητηθεί να γίνουν και κάποιες αποστολές που θα τρέχουν παράλληλα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Ποια είναι η έκταση αυτών των παραλλήλων ασκήσεων. Ε, υπάρχουν κάποιες ε, συγκεκριμένες απαιτήσεις. Μας είπατε για κάποια νούμερα, μας αναφέρατε το 2015. Υπάρχουν κάποια ποσοστά λοιπόν τα οποία θα ισχύουν σε αυτές τις παράλληλες αποστολές. Μετά, ε, έχετε κάποιες συγκεκριμένες προσδοκίες, ε, συγκεκριμένα ε, νούμερα, θέλετε, μας είπατε, αύξηση σε ορισμένους, ορισμένες κατηγορίες. Γιατί αύξηση μιλάμε ακριβώς. Μετά, τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς μας είπατε ότι προς το παρόν δεν θα έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα οι δράσεις. Αναμένετε ή σχεδιάζετε να επεκταθείτε και σε εκτελεστικού χαρακτήρα δράσεις και πότε, σε ποιο, ε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Μετά, άλλη ερώτηση. το πεδίο εφαρμογής, την έκταση που θα καλύψουν αυτές οι δράσεις. Μας είπατε για, κάποιες, ε, για την θαλάσσια ασφάλεια, για μια δράση παγκόσμιας εμβέλειας, για τον, για τον κόλπο της ε, Γουινέας, για το στενό Μαλάκα στην Ινδονησία, για αναπτύξεις ε, δυνάμεων στην θάλασσα της Κίνας. Τι ακριβώς σχεδιάζετε; ποιες είναι οι Απόστολες, σκοπεύετε να στείλετε πολεμικά πλοία εκεί. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα λοιπόν σχέδια γι' αυτό, θα είναι παγκόσμια εμβέλεια η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας είπατε για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων πέραν της ε, επικράτειας του ΝΑΤΟ. Για κάποιες απομακρυσμένες περιοχές μιλήσατε. Τι ακριβώς εννοείτε. Δηλαδή να φανταστώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια για ανάπτυξη δυνάμεων στο στενό Μαλάκα. Τέλος. Βλέπω πως συνεχίζουμε να μιλάμε για την επέκταση ε, της χρηματοδότησης, των τρόπων χρηματοδότησης. Βλέπω ότι στηριζόμαστε όλο ένα και περισσότερο στη σχέση κόστους-όφελους. Αλλά νομίζω πως εδώ είναι κάπως ασαφή τα πράγματα. Κρυβόμαστε πίσω από ρήτρες, από κανόνες. Ε, υπάρχουν όμως κάποια κρατημέλη τα οποία έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν σε κάποιες αποστολές. Νομίζω πως υπάρχουν και αυτά τα κράτη που έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν σε αποστολές θα είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στην χρηματοδότηση αυτών. Είναι δίκοπο μαχαίρι λίγο πιστεύω να μιλάμε από τη μία για επιφυλάξεις, για το ρόλο του Κοινοβουλίου και από την άλλη και ο κύριος Γκάλερ μας μίλησε για ασαφή όρια για θολό τοπίο. Μας είπε ότι δεν έχουμε τα χρήματα, αλλά έχουμε τις δυνατότητες. Αλλά άμα δεν έχουμε τα χρήματα, πώς θα αναπτύξουμε τις ικανότητες και από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για χρήματα τα οποία δεν έχουμε και από πού θα έρθουν, από τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, από ποιους. Και ποιες θα είναι αυτές, οι, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στα δημοσιονομικά μας, ιδιαίτερα για τα οικονομικά αδύναμα κράτη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, Σάμκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να συμμετάσχω και εγώ στη συζήτηση αυτή γιατί έτσι όπω βλέπω εγώ τα πράγματα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την εξή κατάσταση. Τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως τους τελευταίους μήνες, η δουλειά μας στον τομέα της ΚΠΑ έχει επιταχυνθεί πολύ. Οπότε το τρένο έχει μπει σε κίνηση, επιταχύνει. Ωραία. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν ε, με την αρχή του θέματος. Και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ βασικό. Προστιθέμενη αξία. Έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση όπου οι περισσότερες χώρες μέλη είναι μέλη και στο ΝΑΤΟ. Οπότε όλες οι δραστηριότητες τώρα που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, ανταγωνίζονται τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, δρούν συμπληρωματικά τα δύο. Έτσι δεν είναι, πρόκειται για προστιθέμενη αξία, μπορούμε να πούμε. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. αποστολές, στρατιωτικές και μη στρατιωτικές. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις που δεν επιλύονται μόνο με στρατιωτικά μέσα, ούτε μόνο με μη στρατιωτικά μέσα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την τεχνική πρόοδο και την έρευνα. Έχω εκπλαγεί ξανά και ξανά κατά το παρελθόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση έρευνας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Λες και θα μπορούσαμε να έχουμε έρευνα στην συνδεσιμότητα και να την χωρίσουμε στο στρατιωτικό και το μη στρατιωτικό σκέλος. Επιτέλους για πρώτη φορά λοιπόν τώρα έχουμε διαθέσιμα χρήματα, 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, για έρευνα και για να προετοιμάσουμε και πρωτότυπα. Αν λοιπόν έχουμε τα χρήματα αυτά, η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει τι θα ερευνήσουμε, που θα επικεντρωθεί η έρευνά μας και το σύστημα τα πάνη Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων πώς θα έχει. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό και έχω λόγο που το ρωτάω. Γιατί από την δικιά μου εμπειρία τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, αυτά τα προγράμματα δεν έχουν υλοποιηθεί αποτελεσματικά. Πάντα κάτι λείπει, κάτι δεν έχει γίνει σε σχέση με το αρχικό. Οπότε ποιος θα αποφασίσει ποια είναι η προτεραιότητά μας για την έρευνα και ποιος θα είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματικότητα της δαπάνης των κονδυλίων. Δεν είναι δυνατόν να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου στο τέλος τα χρήματα αυτά ή τα περισσότερα χρήματα πηγαίνουν σε δύο ή τρεις οντότητες ή πολυεθνικές στον τομέα της άμυνας. Αν πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια, αυτά θα πρέπει να δαπανώνται πραγματικά αποτελεσματικά. Οπότε εκεί προβλέπετε καμιά λογή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντανζό έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Σερανό. Πράγματι καλύψατε πολύ καλά το θέμα, με φιλοδοξία και πολλά υποσχόμενα. Εγώ δεν είμαι τόσο σαφής στα μπράβο όπως ήταν οι συνάδελφοι, γιατί λέω ότι ναι, οι στόχοι είναι φιλόδοξοι, αλλά παραμένουν στόχοι. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Πολλά ανακοινώνονται, πολλά θετικά, χτες ανακοινώθηκαν πολλά θετικά. Τα χρήματα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι εικονικά προς το παρόν, γιατί πρόκειται για το 2020. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το 2020 πολιτικά μιλώντας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συζήτηση που θα έχουμε για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπω και πολύ καλά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι θα τα βάλουμε αυτά τα χρήματα σε προγράμματα άμυνας, αλλά μέχρι τότε θα γίνουν και εκλογές. Οπότε δεν είμαι σίγουρη ότι για το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να τηρήσει τις υποσχέσεις της, με ό,τι θα κάνει το 2019 δηλαδή. Οπότε εντάξει, πολύ καλή αλλαγή στον προσανατολισμό, αλλά πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Και όλα αυτά τα στοιχεία στο οποία αναφερθήκατε, για άλλη μια φορά πρέπει να ερμηνευτούν και στην πράξη. Οπότε είτε πρόκειται για τις ομάδες μάχης, είτε πρόκειται για την μόνιμα διαρθρωμένη συνεργασία. Εγώ δεν νομίζω ότι προδεύουμε τόσο πολύ. Εντάξει, έχει ανοίξει η συζήτηση. Έτσι κι από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. το ξέρουμε ότι το θέμα αυτό της μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασίας έχει να κάνει με το τι βάζουμε μέσα και τι αφήνουμε απ' έξω. Δεν θέλαμε να την κάνουμε τη συζήτηση, γιατί ξέραμε ότι αυτή θα ήταν η δυσκολία, και όταν την ανοίξαμε την κλείσαμε αμέσω γιατί βρεθήκαμε μπροστά στη δυσκολία. Τώρα ξανανοίξαμε τη συζήτηση, μπράβο, καλά κάναμε, αλλά να βρισκόμαστε απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες. Και προσπαθούμε να βρούμε λύση με ενδιαφέρουσα ορολογία. Αυτό το θέμα το modular inclusivity, ε, δηλαδή ε, μετριασμένη συμπερίληψη, είναι όροι τέλο πάντων που έχουμε εφεύρει και που καταδεικνύουν τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Και το είπε και ο Μικάηλ Γκάλερ πριν από λίγο. Τελικά θα καταλήξουμε σε κάτι ελάχιστο, χωρίς αποκλεισμού, σύμφωνοι, αλλά θα είναι το ελάχιστο και δεν θα έχει τίποτα το διαρθρωμένο και τίποτα το μόνιμο. Γι' αυτό και εγώ δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος για τα όσα λέμε για αυτήν την μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Τα πάτε κι εσείς τι θα γίνει με, τον με την επιχειρησιακή χρηματοδότηση. Νομίζω ότι σωστά λέτε ότι η PSDC τελικά θα εξαρτάται από την ε, επιχείρηση. Αυτή θα είναι η οποία θα σέρνει τα πράγματα. Και πώς θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά στον κόσμο, στους φορολογούμενους. Γιατί όταν μιλάμε για τις ικανότητες χωρίς όμως να έχουμε υπόψη μας και τις επιχειρήσεις, ε, δεν φτάνει. Και το επιχειρησιακό σκέλος υποφέρει από χρηματοδότηση σήμερα. Οπότε για να διευκολύνουμε να κάνουμε να συνεισφέρουν και αυτοί οι οποίοι διστάζουν μέχρι τώρα, αλλά και για να ανακουφίσουμε λίγο αυτούς που συμμετέχουν πολύ, πρέπει να το δούμε αυτό. Αν δεν λύσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό, τότε όλα όσα συζητάμε παραμένουν εικονικά. Άρα επίγει. Είναι πολύ ωραία να υποσχόμαστε πέντε δισεκατομμύρια για μερικά χρόνια, για ικανότητες. Εντάξει, δεν το κάνετε εσείς, η Επιτροπή το κάνει, αλλά εδώ πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της άμεσης χρηματοδότησης. Τέλος. Επανέρχομαι στο όσα ανακοινώθηκαν για τον ε, σχεδιασμό ικανότητας. Πολλά υποσχεθήκαμε εικονικά χρήματα. Αλλά σε ποιο πρόγραμμα θα τα βάλουμε αυτά τα χρήματα. Και πιστεύω ότι εδώ βάζουμε το κάρο πριν από τα ζώα. Πρέπει να καθορίσουμε ποιες θα είναι οι ικανότητες στρατηγικής σημασίας που θα χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι αύριο. Αν αυτό δεν το καθορίσουμε γρήγορα, τότε τα χρήματα, ακόμα αν τα βάλετε το 2020, δεν θα χρησιμεύουν σε τίποτα. Και εκείνοι που θα δυσκολευτούμε όταν θα πρέπει να καθορίσουμε ποιο είναι ο εξοπλισμό ικανότητα στον οποίο θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα. Δεν θα είναι απλό να επιτευχθεί συμφωνία. Και εντάξει, φαντάζομαι ότι θα κατεβάσει τι φιλοδοξίε τη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η συνεργασία θα ξεκινήσει με δύο. Γιατί αν θέλουμε να γίνουμε περισσότερο, θα είναι πιο δύσκολο. Οπότε θέλω να με καταλάβετε καλά. Πρόκειται για σχόλιο βέβαια, όχι τόσο για ερώτηση. Χαίρομαι μεν που υπάρχει αυτή η συνδυτοποίηση που εκφράζεται με δηλώσεις ε, τόσο πρόθυμες λοιπά, Αλλά πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές και ψύχρεμοι γιατί δεν έχουμε φτάσει πουθενά ακόμα. Οπότε θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Πασκού και που το διάβασα κι εγώ. Ότι κάναμε περισσότερα σε δύο χρόνια από ό,τι έχουμε κάνει τα 60 τελευταία. Εμένα με διασκεδάζει γιατί πρώτον δεν ισχύει δεν είναι αλήθεια. Ανακοινώσαμε πολύ περισσότερα σε λίγους μήνες από ό,τι ανακοινώσαμε σε 60 χρόνια. Ναι, αλλά δεν κάναμε περισσότερα στα δύο χρόνια από ό,τι κάναμε στα 60. Και είμαι λίγο νοσταλγικός, τι να κάνουμε, είμαι. Θυμάμαι πως ξεκίνησε η ΠΕΣΔ στις αρχές της δεκαετίας του 90 που είχαν γίνει πολλά. Οπότε να παραμείνουμε ψύχρεμοι απέναντι στις ανακοινώσει που διαδέχονται μία την άλλη τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριο Σοφοζέρ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω αμέσω μετά τον συνάδελφο Ντενζόν. Συγκλίνουν κάποιες απόψει βάσει εθνικότητας, υποθέτω. Λοιπόν, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Άμυνα πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι ποτέ δεν θα υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Και το λέω αυτό γιατί δεν συμμεριζόμαστε, δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις για τον κόσμο μεταξύ μας. Για τη Ρωσία, για παράδειγμα, η Γαλλία δεν βλέπει τη Ρωσία όπως τη βλέπει η Πολωνία ή οι Βαλτικές χώρες. Και αυτή την προσέγγιση μπορούμε να την έχουμε και σε πολλά άλλα στοιχεία που έχουμε να κάνουμε την άμυνα. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και υπογραμμίστηκε Μπορούμε να έχουμε κοινά ε, προγράμματα, μπορούμε να έχουμε και κοινέ δράσεις για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, για παράδειγμα. Οπότε, όταν μιλάμε για διαρθρωμένη συνεργασία, για κοινά σχέδια, κοινέ δράσεις, πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει χρησιμότητα. Να έχουμε δηλαδή τέτοιες δομές συνεργασίας. Βέβαια εδώ μπαίνει το ζήτημα τη συμμετοχής του αποκλεισμού. Αυτό το χαρακτήρα με τη συμμετοχή όλων εγώ δεν βλέπω η συνεργασία πως μπορεί να... Μάλλον πρέπει να προσφέρει προς τα εννοείται από μόνη της. Αν δεν το κάνει πρέπει να σταματήσει. Είναι προφανές. Πρόκειται για συμπληρωματικότητα. Τώρα για την αναθεώρηση. Εγώ θα ήθελα να δουλέψετε πάνω σε αυτά που λείπουν σε μια ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτονομία, κυριαρχία. Χρησιμοποιώ τον όρο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας μερικές φορές. Στην ομάδα μου βέβαια δεν αρέσει και πολύ, πρέπει να προσέχω, τέλος πάντων. Πρέπει να έχουμε μια αυτόνομη ικανότητα ως Ευρωπαίοι για την έρευνα και την ανάπτυξη και την τεχνολογία. Ό,τι έχει να κάνει με την πληροφορική, που είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα και που έχει να κάνει από τα στρατιωτικά... από τα τσίπ ε, κλπ. Αν δεν τα λάβουμε υπόψη μας αυτά, ο στρατός μας δεν θα χρησιμεύει σε τίποτα, γιατί άλλοι έχουν το κλειδί και θα μπορούν να σταματήσουν τα αεροπλάνα μας, τα πλοία μας, να φροντίσουν να μην μπορούν να λειτουργήσουν, τις τηλεπικοινωνίες μας να τα διακόψουν όλα. Οπότε πρέπει συγκεκριμένα να βλέπουμε τα πράγματα με κοινέ δράσεις, κοινά σχέδια που να είναι συμπληρωματικά. Ας αναλύσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση στην αναθεώρηση βάσει του τι λείπει και να προσανατολιστούμε ακριβώς αυτά που μέχρι τώρα λείπουν για να τα καλύψουμε. Για μένα αυτή είναι η στρατηγική που δεν θα είναι ελάχιστη, θα είναι εξαιρετικό αν καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό. Εγώ το πίστεψα το ευρωπαϊκό σχέδιο άμυνας. Το 2000 ήμουνα μόνος. Δύο χώρες πιστεύαν στην εξαρτησία της Ευρώπης, η Γαλλία και η Ρωσία τότε, μόνο. Και ήμασταν μόνοι μας. Κανένας άλλος δεν ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε. Ο κύριος ε, fraud. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρέσβη. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ε, υπάρχει μια κοινή προσέγγιση, βέβαια κάτω από ορισμένου όρου. Ο κ. Ντανζόν ανέφερε του πιο σημαντικού, ότι ωραία όλα αυτά στα χαρτιά, αλλά βεβαίω ε, πρέπει να δούμε και πώς ε, όλα αυτά εν ευθέτω χρόνο θα μπορούσαν να μετατραπούν να γίνουν πραγματικότητα. Μπορεί να συμφωνούμε όλοι ότι η γεωπολιτική κατάσταση ως εξελίσσεται σήμερα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που υπήρχε πριν από 10-15 χρόνια. Διακόπτη πρόεδρος. Όποιος θέλει να φύγει, παρακαλώ να φύγει ήσυχα από την αίθουσα για να μπορούν και άλλοι να λάβουν το λόγο και να μιλήσουν. Λοιπόν, έλεγα Έχουμε τώρα κάποιον στον Λευκό Οίκο που να είναι ε, όσο πιο απρόβλεπτος γίνεται. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά έχουμε έναν προβλέψιμο ε, ηγέτη στη Ρωσία ένα ηγέτη που χρησιμοποιεί τη λογική αλλά και ε, με πάση περιπτώσει η κατάσταση δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί σας λέω, στο Λευκό είχαμε κάποιον άνθρωπο προβλέψιμο που να μπορούμε να τον χειριστούμε. Και έτσι φτάνουμε στο να είμαστε αναγκασμένοι ε, ως Ευρωπαίοι να αντιδράσουμε. Η αντίδρασή μας είναι σήμερα ακόμα πιο σημαντική. Αυτό το μάντρα το οποίο προσπαθώ κάθε φορά να λέω, οποτεδήποτε μου δίνεται ευκαιρία, είναι ότι Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό το έγγραφο που παρουσιάσατε και εσείς και χθε η Κομισιόν, αλλά εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ε, μια κοινή εξωτερική πολιτική με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ε, διαπιστώσαμε ότι στη Συρία αντιδράσαμε μόνο αφού εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων μας χτύπησαν την πόρτα και τότε πια ε, συνειδητοποίησαμε ότι κάτι τρέχει στη γειτονιά μας. Ακόμα και η προσέγγιση του Μίνσκ δεν είναι ευρωπαϊκή, είναι η προσέγγιση δύο ευρωπαϊκών κρατών έναντι της κρίσης που μαστίζει την Ουκρανία εδώ λοιπόν κάτι λείπει. Όμως θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια πράγματα ε, τα οποία αναφέρατε κυρίως σε σχέση με τα battle groups. Γιατί τα battle groups είναι και το πιο συγκεκριμένο, το πιο απτό που έχουμε. Είπατε ότι δέκα ημέρες μετά τη λήψη της απόφασης ότι θα αναπτυχθούν ε, οι μάχημες αυτές τις ομάδες λοιπά. Όμως 10 ημέρες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση μιας κρίσης. Και έτσι φτάνω στο επόμενο ερώτημά μου. Ε, ποιο είναι το κατόφλι για να αναπτυχθούν αυτές οι μάχημες ομάδες. Υπάρχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο σχέδιο το τι θα πρέπει να ε, γίνεται, πώς θα τους δίνεται εντολή ώστε να δραστηριοποιηθούν. Και το τρίτο είναι ε, η κοινή ανάληψη κόστους. Αυτό ε, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος πληρώνει τι και ποιος αντιτίθεται. Τα περισσότερα κρατημέλη αντιτίθενται στο κοινό κόστος. Δεν ξέρω, αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Ε, θα χαιρόμουν να μπορούσατε να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ τον κύριο Φρόιντ. Ε, νομίζω ότι εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ερωτώντων. Ε, θα ήθελα και εγώ να υποβάλω μια ερώτηση, αλλά παρακαλώ να έχετε κατά νου με την ιδιότητά μου του απλού μέλους της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ. Με αυτή λοιπόν την ιδιότητα θα μιλήσω. Καταρχήν να πω ότι από τότε που προτάξα να δουλεύω στην Υποεπιτροπή και από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με τις εξελίξεις ε, στον τομέα της ασφάλειας και της ε, άμυνας. Από τότε λοιπόν διαπίστωσα ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει σύγκληση απόψεων. Κυρίως όσον αφορά τις απειλές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εχθές αυτό που είδα ότι δεν υπήρχε σε αυτά που είπαν η κυρία Μογκερίνη και ο κύριος Κατάινεν, αλλά και σήμερα διαπιστώνω κύριε Πρέσβη, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά Διεπίστωσα ότι δεν υπάρχει ε, σαφής ορισμός ε, των ε, απειλών και των μέτρων που θα κληθούμε να λάβουμε για να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι σε τελική ανάλυση και ο στόχος της ενοποίησης, δηλαδή το να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις ε, απειλές ε, αποτελεσματικότερα. Και όπως ε, έχω πει πολλές φορές, μιλάμε για μια σειρά απειλών σε αντίθεση με αυτά που είχαν προβλεφτεί αρχικά ως στρατηγική μας. Μιλάμε λοιπόν για πολλές απειλές σε πολλές περιοχές, προς Ανατολάς, προς Νότον και όταν μιλάμε για Νότο, ο Νότος ε, διευρύνεται όλο και περισσότερο, δεν φτάνει μέχρι τον Μπαγκλαντές, αλλά όπως σας είπα διευρύνεται η έννοια του Νότου. Ως εκ τούτου, ε, όταν μιλάμε για αυτά τα μέτρα, είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για τις ε, απειλές. Όταν μιλάμε για καλή συνεργασία με το ΝΑΤΟ, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και οι δύο οργανισμοί να μπορούν ε, να χρησιμοποιούν τις δικές τους ε, δυνατότητες για να αντιμετωπιστούν οι απειλές. Αναφερθήκαμε ε, στην υβριδική ε, συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Αλλά εγώ δεν βλέπω να υπάρχουν τέτοιου είδου μέτρα. Εκτός από το υβριδικό κέντρο, το οποίο δημιουργήθηκε πρόσφατα στη Φινλανδία και που εμείς θα το στηρίξουμε είναι το μόνο, το ευρυδικό κέντρο για το οποίο γίνεται συγκεκριμένα λόγος. Και Ξεκολουθούμε όμως να μην ονοματίζουμε τη χώρα η οποία απειλεί την ασφάλειά μας ε, και όταν γίνεται και λόγος για την υβριδική μορφή, κατ' ουσίαν αναφερόμαστε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη Μολδαβία. Όσον αφορά τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Ρωσία είναι πολύ σημαντική στην περίπτωση αυτή ε, για να λύσουμε τα προβλήματα ασφάλειας της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Διερωτώ με λοιπόν κατά πόσον αυτό ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με μια χώρα η οποία όμως παράλληλα σε επίπεδο εμπειριδικό αποτελεί και απειλή. Δεν εξετάζουμε το θέμα της Ουκρανίας ή της Γεωργίας παρότι και οι δύο χώρες ε, ε, καταβάλουν προσπάθειες ε, στους κόλπους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν τους έχουμε επιλέξει ως συνεργάτες στην ανάπτυξη των προσπαθειών μας. Την Ισία, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά τι γίνεται με την Ανατολική Μεσόγειο και με την ε, αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Η σταθεροποίηση της ετηνησίας είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορούν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις ε, του ΝΑΤΟ, δηλαδή οι επιχειρήσεις ε, του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και όλες οι άλλες θαλάσσιες επιχειρήσεις. Διερωτώμε λοιπόν κατά πόσον ε, θα πρέπει να κατονομάσουμε ίσως και άλλους εταίρους. Έχω αρκετά ερωτήματα που αφορούν στην ΠΕΣΚΟ. Ίσως ε, κύριε Πρέσβη μπορείτε να μας ε, εξηγήσετε ποια είναι τα μεμονωμένα κράτη, η θέση των κρατών που αφορούν στην ΠΕΣΚΟ. Και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η ΠΕΣΚΟ, διότι έχουμε ένα πακέτο δέσμη μέτρων ε, αμυντικού χαρακτήρα και εκεί προφανώς και παίζει ρόλο το στοιχείο βιομηχανία. Θεωρώ ότι η συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθοριστικής ε, σημασίας. Όσον αφορά το βιομηχανικό σκέλος, Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα περιστούν οι οικονομίες κλίμακος ε, τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή. Και όταν μιλάμε για την άμυνα, όταν μιλάμε για θαλάσσιες επιχειρήσεις, νομίζω ότι είναι δύσκολο ακόμα και να φανταστούμε την έλλειψη συνεργασίας έλλειψη συνεργασίας με ένα σημαντικό ή με κάποια σημαντικά ε, θαλάσσια κράτη για να πετύχουν οι θαλάσσιες επιχείρησεις, όπως είναι η επιχείρηση Αταλάντα. Υπάρχει το θέμα της εμπειρίας που μπορούμε να κερδίσουμε από τη συνεργασία με την ναυτιλία Αυτό είναι ένα θέμα σε πάρα πολλούς τομείς. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο και για να τη χρησιμοποιήσουμε και για αποτροπή, εκφοβισμό σε σχέση με απειλές που αντιμετωπίζουμε. Παρότι λοιπόν κατανοώ τη σκληρή δουλειά που γίνεται στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και εδώ παίζει σίγουρα ρόλο η Κομισιόν Όλα αυτά συμπίπτουν με τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης συμπίπτουν και με την έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων για το Brexit. Φαίνεται ότι αυτό που χρειάζεται είναι να ακούσουμε το ανώτατο όριο, το τι μπορεί να προκύψει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Γιατί έχουμε ακούσει επανειλημμένα ότι τώρα είμαστε πρόθυμοι να ε, προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να υποβάλουμε ερωτήσεις ε, και πρέπει να ρωτήσουμε πώς πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι ικανότητες που είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολύ σημαντικές ε, για την Ευρώπη, και σε επίπεδο πληροφορικής και εδώ αναφέρουμε σε αυτά που είπε ο κ. Σαφχάουζεν. Θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα με την ανάπτυξη των battle groups. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα που συζητήσαμε προηγουμένως του Ανατολικού Κονγκό. Ξέρουμε ότι υπήρχε, υπάρχει πλέον μικρότερη συνεργασία ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις του Κονγκό και αυτές του Βελγίου. Και γι' αυτό λοιπόν διαρωτώ Θα στηρίξουμε κι εμείς ε, την προστασία των συνόρων της Ουκρανίας. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Αυτό είπε ο κύριος Σαφχάουζεν αλλά κατ' ουσίαν κανείς δεν μίλησε για τις ε, απειλές και για την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές. Εξακολουθούμε να μιλάμε για συνεργασία και για ολοκλήρωση, ίσως ε, και για ευρωπαϊκή αυτονομία και πολύ συχνά επαναλαμβάνεται ε, και λόγω ίσως της απομόνωσης της Αμερικής. προφανώς και απορρέουν απειλές από αυτόν τον απομονωτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν το βλέπουμε. Ας πούμε στη δική μου την περιοχή ε, εξακολουθούν να υπάρχουν ε, αμερικανικά στρατεύματα. Ως εκ τούτου ε, θα πρέπει να συζητήσουμε για μια σειρά πολιτικών θεμάτων. Παρακαλώ κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Um, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για τη συνεισφορά σας στην συζήτηση. Ευχαριστώ όλους εσάς, ευρωβουλευτές, για τα σχόλια, για τους προβληματισμούς που εκφράσατε, για τη στήριξη, για τα ενθαρρυντικά σας λόγια, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Να καταστήσω σαφές ότι έχουμε απόλυτη επίγνωση του ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Η Αντιπρόεδρος Μογκερίνη πρέπει να σας πω ότι έχει δηλώσει τη δέσμευσή της για αυτή την ατζέντα και υπάρχουν πολλά έργα τα οποία δρομολογούνται. Δεν δρομολογούνται όμως ε, ακόμα. Πρέπει να γίνει αυτό για να φτάσουμε στην εφαρμογή. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα ενδιάμεσο στάδιο που έχουν γίνει πολλά, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν ακόμα περισσότερα έτσι ώστε να καρποφορήσουν οι προσπάθειές μας και να δούμε πραγματικά αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν να ε, ασχοληθούμε με τη δρομολόγηση των προγραμμάτων που πρέπει να ξεκινήσουν. Διαφορετικά δεν θα φτάσουμε στο επόμενο στάδιο. Είναι λοιπόν, πιστεύω, απλή λογική. Αναφερθήκατε σε απειλές Και έχετε δίκιο. Συνήθως οι παρουσιάσεις μου αφορούν και τις απειλές. Το έκανα για οικονομία χρόνου, αν θέλετε, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Η ύπαρξη αποτελεσματικών δομών και ύπαρξη ικανοτήτων έχουν νόημα μόνο αν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Αλλά γιατί γίνεται τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή και γιατί είναι σύμπτωση αυτή. Γιατί αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει έτσι μία τόνωση του αμυντικού εξοπλισμού. Δεν είναι καθόλου σύμπτωση. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν δεδομένα που, έχουν, που δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πληγεί σε θέματα ασφαλείας και χωρίς ενίσχυση της ασφάλειας δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε ε, τις ελλείψεις μας όπως πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν πιέζουμε για μεταρρυθμίσεις, γι' αυτό λοιπόν αναλαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε. Ε, υπάρχουν απειλές ε, στα ανατολικά, στη Μέση Ανατολή και υπάρχουν απειλές στα νότια. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συγκεντρώνονται και δημιουργούν μία άτυχη συγκυρία, διότι έχουμε απειλές ε, σε, ολούθε σε όλη την γειτονία της Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ε, ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν ικανότητα άμυνας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην ξεχνάμε, έχει διαφορετικό ρόλο από ότι το ΝΑΤΟ. Έχει ε, τον ρόλο της διασφάλισης ασφάλειας μέσω αμυντικών μέσων, μέσω των ε, μέσων διαχείρισης κρίσεων που έχουμε και αυτά είναι δεδομένα επίσης έχει και δυνατότητες που δεν τις έχει το ΝΑΤΟ. Διπλωματική δυνατότητα, ε, έχει και τη δυνατότητα μέσω της οικονομικής συνεργασίας, μέσω του εμπορίου να ασκήσει πίεση και να αλλάξει ε, πράγματα. Δεν λοιπόν αυξάνει την ασφάλεια μόνο μέσω της άμυνας, αλλά χρειάζεται και αυτή η άμυνα εάν θέλεις να σε ε, πάνω στα σοβαρά και αν θέλεις να αντιμετωπίσεις επιτυχώς τις εξωτερικές επιλές. Ελπίζω λοιπόν ε, να καταλάβατε ε, τώρα. Ελπίζω να κατάφερα να αντιμετωπίσω να απαντήσω στα σχόλιά σας, στα επικριτικά σας σχόλια και να είστε σίγουροι ότι ε, δεν φταίει η πολιτική μας, αλλά ίσως έφταγε η παρουσίασή μου που ε, δεν συμπεριέλαβε και αυτό το θέμα. Με τα χαράς λοιπόν να σας εξηγήσω και προσωπικά τι γίνεται ακριβώς με τις δράσεις, σε ποια παιδεία, ποιες περιοχές δραστηριοποιούμαστε. Με τα χαράς λοιπόν και σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τώρα αναφέρθηκαν και άλλα για το NPCC, την στρατιωτη, τις στρατιωτικές ικανότητες, αν θα περάσουν σε στάδιο εκτέλεσης ή όχι. Ε, εντάξει, νομίζω πως είναι ένα ερώτημα που ορθώς ε, θέσατε. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Προβλέπετε μία αναθεώρηση για το 2018 και τότε θα είναι σημαντικό να δούμε πόσο αποτελεσματικές ήταν αυτές οι δομές τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Νομίζω πως ήδη έχουμε δώσει μια πρώτη γεύση στα κράτη-μέλη για το τι μπορούμε να επιτύχουμε από τις Βρυξέλλες σε τέτοιες ε, αποστολές και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σύστημα διοίκησης των διαφορών επιχειρήσεων, υπάρχουν διάφορα ε, κεντρικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Northwood, όπως είπατε και εσείς πρόεδρε, στο Ενωμένο Βασίλειο, στο Παρίσι, όπου, από όπου μπορούμε να ε, ελέγξουμε και να αναπτύξουμε αυτά τα έργα. Στο Βερολίνο, στο Πότσταμ υπάρχουν λοιπόν κέντρα. Ε, υπάρχουν, υπάρχει και η συμφωνία ε, Βερολίνο Plus Η επιχείρηση Αλθία στη Βοσνία Τσεκοβίνη επίσης ήταν μια κοινή επιχείρηση. Τώρα, εάν χρειάζεται μια κοινή δομή ή όχι, δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω. Τα κρατη είναι αρμόδια για να απαντήσουν αυτή την ερώτηση, όμως ε, θα το συζητήσουμε και στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχόλια του κυρίου Γκάλερ για την ΠΕΣΚΟ και την ΠΕΠΚΟ μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε και νομίζω πως ε, όντως έχετε ένα πολύ ε, σωστό επιχείρημα. Δεν πρέπει να ε, να περάσουμε στην ΠΕΠΚΟ αλλά στην ΠΕΣΚΟ και αυτό θα πρέπει να είναι μια προειδοποίηση για όλους. Και πιστεύω πως πρέπει να ανοίξει επιτέλους η κουβέντα για το τι αποτελέσματα έχει ε, φέρει η ΠΕΠΚΟ. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Ελπίζω να κλείσει επιτυχώς. Βέβαια πρέπει να καταλάβετε πως υπάρχουν πολλοί αρμόδιοι. Είναι και δικό μας έργο να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε με ιδέες, με προτάσεις ε, και με την ταυτοποίηση, και, ε, ε, ταυτοποίηση σημείων σύγκλησης, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την διαμόρφωση άποψης. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για να ε, επιτύχουμε το στόχο μας και να προσπαθήσουμε τα κράτη-μέλη που έχουν δείξει φιλοδοξία και έχουν φιλοδοξίες προτάσεις να τα προωθήσουμε, χωρίς όμως να μείνουν πίσω άλλοι. Δεν πρέπει κανένα κράτος μέλος να αισθάνεται παραμελημένο. Αυτό είναι και ο θεσμικός μας ρόλος άλλωστε, αλλά είναι επίσης και προς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη. Μπορούμε με διάφορους τρόπους να το επιτύχουμε αυτό στην προκειμένη ή με τον τρόπο που συζητούμε για το πώς πρέπει να είναι η ΠΕΣΚΟ. Αν δείτε τις συνθήκες, αναφέρονται σε λίγα κράτη-μέλη που μπορούν από κοινού να στείλουν μια κοινοποίηση και να ζητήσουν τη συνέχεια μέσω ε, ειδικής πλειοψηφία. Όμως εμείς προσπαθούμε να έχουμε μία εις συζήτηση για το πώς θα είναι δομημένη η ΠΕΣΚΟ. Και σε ό,τι αφορά τα διάφορα έργα, αυτά συνδέονται άμεσα με τα σχέδια ικανοτήτων που αναθεωρούμε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας μας σε παγκόσμιο πλαίσιο και προσπαθούμε δεδομένης αυτής της φιλοδοξίας που θέλουμε να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που θέλουμε και τι είναι αυτό που θέλουμε να αναπτύξουμε από κοινού. Έτσι ώστε να μην ωφελήσει μόνο την αμυντική βιομηχανία, να, αλλά να δημιουργήσει και οικονομίες κλίμακας, να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την τεχνολογική και ερευνητική πρωτιά, την οποία δεν θα διατηρήσουμε αν ο καθένα είναι απομονωμένο και εργάζεται μόνος του. Βλέπετε λοιπόν ότι τα ωφέλη είναι πολλά. Και μαζί με τα κράτη-μέλη προσπαθούμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα με ρωτήσατε ποιο κράτος μέλος είναι, πού, τι ακριβώς γίνεται. Νομίζω πως ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται, ποια κράτη-μέλη έχουν δείξει περισσότερο ενθουσιασμό και ποια όχι να πω ότι η Αντιπρόεδρος Μοκερίνη πάλι αναφέρθηκε στο θέμα της ΠΕΣΚΟ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτός ο σκεπτικισμός αφορά περισσότερο το πόσο πρόθυμοι είμαστε να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Και στην πρώτη συνάντηση που είχαμε θέμα την ΠΕΣΚΟ με τους διευθυντές αμυντικής πολιτικής είδα ότι όλοι πλέον γνωρίζουν ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε και το ερώτημα που τους απασχολεί είναι το πώς. Αυτά σε ό,τι αφορά την φιλοδοξία μας. Όμως νομίζω πως όλοι θέλουν να υπάρξει συνέχεια και πρόοδος. Μετά, ποιος θα συμμετέχει στην ΠΕΣΚΟ. Νομίζω πως είναι προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξει κάποιες θέσεις σε μη μέλη, σε τρίτες χώρες. Εάν υπάρχουν κάποια τρίτα μέλη που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη διαφόρων έργων, θεωρώ πως αυτό είναι ένα πολύ θετικό. Και αυτό συζητιέται λοιπόν ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Τι άλλο με ρωτήσατε. η ε, συμμετοχή. σε κάποιο έργο, σε κάποιο project, αν αυτό δίνει δικαιώματα ψήφου. Κύριε Πάσκορο, το ρωτήσατε νομίζω εσεί αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο και πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει αποδοχή των κοινών δεσμεύσεων. Αυτό μπορεί να είναι τα επίπεδα επενδύσεων, Μπορεί να είναι η συμμετοχή σε διάφορα κοινά project, μπορεί να είναι η συμμετοχή σε διάφορες επιχειρήσεις. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Πρέπει λοιπόν να θεσπιστούν κάποια όρια ή τουλάχιστον να υπάρχει μια δέσμευση από τα κράτη-μέλη για έναν ευρύτερο ε, στόχο. Και μετά από αυτό να περάσουμε στη συνέχεια στα επιμέρους έργα που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Αυτές οι κοινέ δεσμεύσεις πρέπει να οδηγήσουν και σε μεγαλύτερη συνοχή και σε συνεργασία. Συνεργασία, όπως είπατε κι εσείς, και όχι συντονισμό. Τώρα, ω κράτο μέλος πρέπει πρώτα να αναλάβετε δεσμεύσεις και μετά να αναλάβετε κάποιο project. Πρώτα λοιπόν έρχονται οι δεσμεύσεις οι οποίες σας δίνουν και το δικαίωμα ψήφου. ψήφου σε αυτά τα projects στα οποία συμμετέχετε. Εάν ας πούμε υπάρχει κάτι που τρέχουν άλλα κρατημέλη, εσείς δεν μπορείτε να ψηφίσετε αν έχετε αποφασίσει να μην συμμετέχετε σε αυτό. Τώρα περνάμε όλοι σε ένα άλλο στάδιο, όπως είπατε κύριε Πάσκο, ανάπτυξης δυνάμεων. Κοιτάξτε, χρειάζεται να περάσουμε σε αυτό το σχέδιο, χρειάζεται να υπάρχουν τέτοιες ε, δυνάμεις. Υπάρχουν, υπάρχει αυτή η αναγνώριση από πολλά κράτη-μέλη, όπως ε, όλοι γνωρίζουν ότι πρέπει να αναπτύξουμε ικανότητες. Υπάρχει και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σχετικά. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ειδικευτεί στις ε, λεπτομέρειες της ε, ανάπτυξης αυτών των δυνάμεων. Γιατί μέλημά μας είναι και η προστασία της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αναπτύξουμε εσωτερικά διάφορους ε, τρόπους άμυνας της Ευρώπης. Η Frontex συμμετέχει ενεργά σε αυτό και τα ερχόμενα χρόνια θα γίνουν πολλά περισσότερα. Ένα παράδειγμα μόνο. Η Λιβύη. Βλέπουμε μια θαλάσσια επιχείρηση σύμφωνα την επιχείρηση Σοφία στα πλαίσια της ε, ΚΙΠΑ και υπάρχει και μια θαλάσσια επιχείρηση στο Βορρά. Αυτή είναι μια συνεργασία εσωτερικών και εξωτερικών μέσων για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Κινούνται λοιπόν τα πράγματα. Και να επιστρέψω και στην ερώτηση της κυρίας Λόζιν για την θαλάσσια παρουσία μας. Οι δύο επιχειρήσεις που έχουμε αναπτύξει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην ακτή της Ομαλίας καλύπτουν πολύ σημαντικές περιοχές, σημαντικές για την ασφάλεια την Ευρώπη και για την θαλάσσια ασφάλεια. Και η εντολή των επιχειρήσεων αυτών μπορεί να είναι βέβαια κάπως περιορισμένη, συγκεκριμένα εκείνη στην ακτή της Ομαλίας, αλλά ε, το έργο τους είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί διασφαλίζει την ε, ασφάλεια ακριβώς ε, μόνο της παρουσίας του εκεί. Και προβλέπονται λοιπόν περισσότερα περισσότερες λεπτομέρειες αυτό το έγγραφο προβληματισμού που θα ακολουθήσει την Λευκή Βίβλο. Τι δηλαδή θέλει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από, σχετικά με την παρουσία της στη θάλασσα. Πού, κεντρική Μεσόγειο, ακτή της Ομαλίας, νοτιοανατολική... Ε, χρειάζεται η Ευρώπη λοιπόν να έχει ασφάλεια. Τώρα αν αυτή η ασφάλεια θα αναπτυχθεί στα σύνορα ή εκτός αυτών, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσουν στα κράτη-μέλη. Και το θέμα της ακτής της Γουινέας είναι κάτι τελείως διαφορετικό παρεπιπτόντος. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω πως ε, σε ό,τι αυτό θα συνεχίσει να ε, έχει μια παρουσία εκεί για πολλά χρόνια. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, και πολλές άλλες ε, ερωτήσεις, απλά προσπαθώ λιγάκι στα χαρτιά μου να δω. Ε, νομίζω ότι έθιξα τα περισσότερα θέματα. Όσον αφορά την κοινή ανάληψη κόστους και τις, τα battle groups, βεβαίως και θα χαρούμε πάρα πολύ αν τελικά μας υποστηρίξετε. Νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκα πλήρως το χρόνο μου. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σήμερα το πρωί και εμείς στη διάθεσή σας. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και εμείς ε, για όλα αυτά που μας είπατε. Δίχως άλλο, ήταν ε, μια πολύ επικατομητική, ενημερωτική συνάντηση. Πιστεύω όμως πως χρειαζόμαστε ακόμα την παρουσία σας περισσότερο για να συζητήσουμε αυτά που θίξατε ήδη. Τη σχέση δηλαδή ανάμεσα στην πληθώρα των μέτρων, τις τακτικές απειλές και τι είδους δράσεις θα αναλάβουμε στους διάφορους χώρους επιχειρήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Thank Please stay. Παρακαλώ, παραμείνετε στην αίθουσα, γιατί έχουμε ακόμα σημαντικά θέματα. Το ένα είναι η ενημέρωση σχετικά με την Αρινή Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα στην Τυφλίδα. Η κυρία Βακαηλή, που είναι πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας, θα έρθει χωρίς άλλη καθυστέρηση. Σας δίνω και το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έλαβε χώρα στην Τυφλίδα, στη Γεωργία, 26 με 29 Μαΐου. Ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια που οργανώθηκε τέτοια συνάντηση σε χώρα μη μέλος της συμμαχίας. Και φάνηκε έτσι πόσο ενδιαφέρεται για το ΝΑΤΟ Γεωργία, όπως επίσης το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ να έχει ομάδες μάχη με άλλες χώρες εκτός ΝΑΤΟ. Ήμασταν τέσσερις. Ο κύριος Χόνος από τους Σοσιαλιστές, Κρεζοτεύσκη από το ECR και ο κύριος Ράντος από την Άλντε. Δύο πράγματα θα ήθελα να υπογραμμίσω. Το ένα είναι τα βασικά που συζητήσαμε στις διάφορες επιτροπές ε, και στην Ολομέλεια αλλά και διμερός. Για την ε, συνέλευση ήταν ενημερωτική συνάντηση, κυρίως όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΝΑΤΟ, που ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκε. Λίγες μέρες μετά τη συνάντηση των ηγετών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Η συνεργασία αυτή λοιπόν βρέθηκε ως προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη και της Ολομέλειας, αλλά και των άλλων επαφών αναφέρθηκαν οι προκλήσεις και για πρώτη φορά είχε τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρει ουσιοδός σε μία έκθεση του ΝΑΤΟ. Ελήφθησαν υπόψη λοιπόν οι θέσεις μας από τον εισηγητή. Το κείμενό μας εκτιμήθηκε πολύ και οι θέσεις μας και ήταν και συνάφθησε το κείμενο. Επίσης, το θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης, της βιομηχανικής βάσης, αλλά και η πρόταση που περιμέναμε της Επιτροπής για κονδύλια στην άμυνα εγκρίθηκαν και συζητήθηκαν και σε δύο άλλες επιτροπές. Επιπλέον, επικεντρωθήκαμε στο ρόλο της συμμαχίας στο Αφγανιστάν, η ε, επιπτώση της κλιματικής αλλαγής, γεωπολιτικές επίσης στην Αρκτική, αλλά και επιπτώσεις των μέσων ε, κοινωνικής δικτύωσης. Φυσικά θέμα ήταν εκεί η Συρία. Πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας. Συστήθηκε το θέμα λοιπόν με τη Ρωσία. Υπήρξε και δήλωση που εγκρίθηκε για την ε, ευρωατλαντική ένταξη της Γεωργίας. Και στην Ολομέλεια υπουργό της Γεωργία, μίλησε για ένταξη τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αναπληρωτής των Γενικών Γραμματέα του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στα εξή. Στη συνάντηση των ηγετών του ΝΑΤΟ την 25η Μαΐου στις Βρυξέλλες και στο ρόλο του ΝΑΤΟ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως επίσης και την κατανομή των βαρών, την ισότιμη κατανομή των βαρών μεταξύ των μελών. Ε, κύριε Γκέτε Μίλλερ προσπάθησε να καθησυχάσει τους συμμετέχοντες για τις Ηνωμένε Πολιτείε, για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που θα στηρίξει το άρθρο 5, είπε. Ίσως υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες μετά τη συνάντηση των 7, αλλά ήταν καθησυχαστικό και η συνεργασία ή πενά το Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ζήτησε από τους βουλευτές να ενθαρρύνουν την στρατηγική εταιρική σχέση. Γιατί ρωτήσαμε επίσης για το πώς βλέπουν οι βουλευτές την ε, συνεργασία αυτή, απάντησε πολύ θετικά και ζήτησε να κάνουμε και εμείς περισσότερες προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας αυτής. Τέλος, οι τρεις διμερείς συναντήσεις που οργανώθηκαν ήταν μια πολύ σημαντική με πολύ καλή ενημέρωση από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας στη Γεωργία, γιατί έχουμε τέτοια εκεί, και ο πρέσβης Γιακάσκος μας ενημέρωσε για τις ε, εποπτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε η μόνη διεθνής παρουσία εκεί και μας ενημέρωσε και για τις δραστηριότητες στην ε, οριακή γραμμή. Η κατάσταση είναι σταθερή προς το παρόν και είπε ότι πιστεύει πως η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γι' αυτό. Γιατί είναι κάτι που σέβονται και δύο πλευρές, και η Ρωσική και εκείνη της Γεωργίας. Μια άλλη συνάντηση ήταν με τρία μέλη από την αντιπροσωπεία του Μαυροβουνίου για την προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συμμαχία. Συζητήσαμε την κατάσταση ασφάλειας στη χώρα και στα Δυτικά Βαλκάνια γενικότερα και ενημερωθήκαμε για την εσωτερική κατάσταση, όπως επίσης και για τις έρευνες που συνεχίζονται μετά τις υπόνοιες για απόπειρα πραξικοπήματος την ημέρα των εκλογών στο Μαυροβούνιο και ενδεχομένως την εμπλοκή της Ρωσίας. Στη συνάντησή μου λοιπόν με τον κύριο Παολάλη, ε, που ήταν και εκείνος που οργάνωσε αυτή τη συνάντηση, συμφωνήσαμε ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι διοργανικές σχέσεις, κυρίως όσον αφορά τις ε, κοινέ εκδηλώσεις στο μέλλον και επίσης συμφωνήσαμε ότι πρέπει να βελτιωθεί ο ρόλος ε, και οι δυνατότητες ε, του ΔΙΝΑΤ μέσα στη συνέλευση να προάγουμε γενικότερα τη συνεργασία στο ΝΑΤΟ. Θα ήθελα επίσης να σε ενημερώσω ότι επιτόπου μπορέσαμε στη Γεωργία να επισκεφτούμε την συνοριακή γραμμή που είναι κοντά στην Νότιο Σετία. Ε, μας παρουσίασαν την ε, προοπτική, την άποψη της Γεωργίας για την κατάσταση. Ε, και βεβαίως συμμετείχαμε ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να υπάρξει συνέχιση και συμφωνήσαμε ότι με τον κύριο Άλλη θα συνδιοργανώσουμε το DNAT, ένα κοινό σεμινάριο προς το τέλος του έτους, σεμινάριο υψηλού επίπεδου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αργότερα θα ορίσουμε τα συγκεκριμένα θέματα. Και θα στείλουμε προσκλήσεις στον κύριο Ταγιάννη, στον κύριο Στόλτενμπερκ, και στην κυρία Μογκερίνη. Με αυτήν λοιπόν την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι θα υπάρξουν και συναντήσεις και επιτόπου επισκέψεις ε, στο ΝΑΤΟ ε, στις Βρυξέλλες ε, πρέπει να παρακολουθήσουμε και την έκθεση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ελπίζουμε αυτό να εγκριθεί στην επόμενη συνάντηση στο Βουκουρέστι 6 έως 9 Οκτωβρίου. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε, για αυτή την ε, ενημερωτική παρουσίαση σχετικά με την συνάντηση ε, ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ και της κοινοβουλευτικής μας συνέλευσης στην Τυφλίδα. Νομίζω δύο φορές ήρθε εδώ στις Βρυξέλλες η ε, εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τυφλίδα και υπήρξε επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Γεωργίας ε, κοντά στα σύνορα, άρα δηλαδή επισκέψει και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι είναι μόνιμη η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την αντιπροσωπεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα άλλο αίτημα να αναλάβει κανείς ε, το λόγο για αυτό το θέμα. Ε, θα ήθελα τώρα να αρχίσουμε την ενημέρωση για την Ιαπωνία. Όμως λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για την ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, που θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω ότι ήταν καλύτερα το θέμα αυτό να το αναβάλουμε για την επόμενη συνάντησή μας. Και απλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι η αποστολή της Επιτροπής μας ε, στην Ιαπωνία ήταν πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολλοί από όσους συμμετείχαν ε, θεωρούν ότι σημειώσαμε και μεγάλη επιτυχία. Μπορέσαμε να συνδυθούμε με στελέχη υψηλού επίπεδου με την ε, κυβέρνηση της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένου ε, του Υπουργού Εξωτερικών, Υπουργός ε, Κίση. Είναι ο αδελφός του Πρωθυπουργού. Και συναντηθήκαμε και με τον ε, Γενικό Γραμματέα για θέματα άμυνας. Επίσης, συναντηθήκαμε με διακεκριμένους βουλευτές συμπεριλαμβανομένου ε, και του κύριο Σιχάρα που νομίζω είναι ο πρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής Φιλίας ανάμεσα στην Ιαπωνία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. βάση το Σύνταγμα της Ιαπωνίας δεν, ε, δεν υπάρχει μόνο άμυνα, αλλά και self-defense, άμυνα Στο Τόκιο υπάρχει ε, ένα ναυπηγείο στη Γιοκοχάμα. Και είδαμε εκεί σκάφη που ναυπηγούνται και ε, σκάφη ακτοφυλακής αλλά και παγοτραυστικά για κάποιες ε, ειδικέ επιχειρήσεις. Είχαμε επίσης τη δυνατότητα να επισκεφτούμε την ναυτική βάση της Γιοκοσούκα και να συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς ασφάλειας, άμυνας, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ιαπωνική άμυνα. συναντήσαμε και τον ε, επικεφαλής ε, της ε, αμυντικής ναυτικής δύναμης της Ιαπωνίας και επισκεφθήκαμε επίσης και ένα πολεμικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο σε αυτή τη βάση. Επίσης συναντηθήκαμε με διάφορα υψηλόβαθμα ε, στελέχη της Ιαπωνίας ε, του Υπουργείου Άμυνα. Είχαμε μία αρκετά πλήρη ενημέρωση για τις εξωτερικές απειλές, όχι μόνο κοντινές, και αποκτήσαμε νομίζω μία πλήρη εικόνα σχετικά με τις ε, απειλές που αντιμετωπίζει η Ιαπωνία στις ε, θαλάσσιες ε, πορευματικές οδούς που τη συνδέουν με την Ευρώπη, στην Ανατολική Κινέζικη θάλασσα. Για παράδειγμα, ήταν ιδιαίτερα έντονες επίσης οι ανησυχίες τους για την απειλή της Βόρειας Κορέας και αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είχαμε. Γι' αυτό λοιπόν επιτρέψτε μου να αναβάλω την ε, ενημέρωση για την επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας και νομίζω πως αν δεν έχουμε κάτι στα διάφορα που δεν το βλέπω τότε θα σας ενημερώσω ότι στις 21 και 22 Ιουνίου θα είναι οι επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Η μερίσια διέταξη για τότε είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ευρωβουλευτές για τη σημαντική συνεισφορά τους, να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων και να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ πολύ.